Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε να αρχίσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχει βαρύ πρόγραμμα και τις δύο ημέρες. Πάμε στο σημείο 1, την έκθεση του κυρίου Ρώση για τα μέτρα προστασίας από τα σε επιβλαβείς, ε, επιβλαβείς οργανισμούς της ουσίας να το βάλουμε ε, πιο μπροστά αντί για τη φάρμακο επαγρύπνηση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εντάξει, έτσι θα γίνει. Προχωρούμε. Σημείο 2. Όλες τις γλώσσες έχουμε εκτός από εστονικά και μαλτέζικα. Δεύτερη ανακοίνωση. Η εβδομάδα Mind Your Heart, φροντίδα της καρδιάς, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου απόψε υπάρχει μια εκδήλωση από τις 7 μέχρι τις 8 με θα έρθει και ο Επίτροπος Μπόρκ ε, και ο Λιθουανός Υπουργός Υγείας επίσης και ο κύριος Μπερτολίνη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και όλα αυτά θα γίνουν στις 7 το βράδυ. Και η ομάδα του Elk Heart Group κάνει αυτό. Η Λίντα Μακέβαν και ο συνάδελφος Παρτανόβα θα προεδρεύσουν. υπάρχει και στο φακελό σας. Έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών εδώ παρούσα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πού είναι, δεν τους βλέπω όμως, δεν έχουν έρθει ακόμα. Ήρθαν ε, από το Υπουργείο Ενέργειας και Αλλαγής Κλίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Α, θα έρθουν στις 4.30. Επίσης, κάποιοι τριμερείς διάλογοι ε, πρέπει να προετοιμαστούν. Ο δεύτερος ε, για το AVS από τη συνάδελφο Σαντρίτ Μπελιέ στις 5 Νοεμβρίου στις 2.30 το μεσημέρι θα γίνει. Μετά έχουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, νομοθετική διαδικασία. Αυτό το επεξεργάζεται ο συνάδελφος μου 5 Νοεμβρίου επίσης και το Sound Level of Motor Vehicles, η έκθεση του κυρίου Ούτσκι για το θόρυβο που κάνουν τα μηχανοκίνητα οχήματα ή ο τριμερής διάλογος που και αυτός θα γίνει 5 Νοεμβρίου. Και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι είναι παρόντες. Συνεχίζουμε λοιπόν και έχουμε και φορτωμένο πρόγραμμα. Αύριο θα συναντηθούμε για το θέμα των αυτοκινήτων με την Προεδρία του Συμβουλίου και θα συζητήσω με τη συνέχεια θα δοθεί με την σημαντική αυτή νομοθεσία για το διοξίδιο του άνθρακα και τα αυτοκίνητα και τις κλινικές δοκιμές, clinical trials. Εδώ θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου ο πρώτος διάλογος και ο δεύτερος έχει προγραμματιστεί για 13 Νοεμβρίου. Ε, για τα f 4 Νοεμβρίου από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι λοιπόν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα με τους τριμερείς διαλόγους και τις επόμενες εβδομάδες ο φόρτος εργασίας δεν θα μειωθεί. Προχωρούμε στο σημείο 3 έγκριση των πρακτικών 29-30 Μαΐου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Και πάμε τώρα στο σημείο 4. Ανταλλαγή απόψε με τον Γκουίντο Ράζη, εκτελεστικό διευθυντή του ΕΜΑ. Ε, εμείς ενημερωνόμαστε πολύ, έχουμε πολύ καλή επαφή με τον οργανισμό και βεβαίως μας βοηθάει και η Dagmar Roth που είναι πολύ δραστήρια και έχουμε συνεχής ανταλλαγής απόψεων. Και Έχουμε λάβει πολλές αποφάσεις στην περίοδο αυτή για τις κλινικές δοκιμές που προανέφερα, την έκθεση της ίδιας της Ντάγμαροτ Μπέρν για τα ιατρικά μηχανήματα, για τεχνολογικά προϊόντα, που δημιούργησε πολλές αντιπαραθέσεις και διαφορετικές απόψεις ε, εδώ στην Επιτροπή και έχουμε και το θέμα της απαλλαγής που μας απασχόλησε πολύ. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση τώρα και να μιλάμε περισσότερο μεταξύ μας, όχι ο ένας για τον άλλο, γιατί ε, δεν ήταν και πολύ ωραία αυτά που έγιναν. Ελπίζω να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον. Πήγαμε πρόσφατα, το πρώτο εξάμεινο δηλαδή, στο Λονδίνο. Η προετοιμασία έγινε από την κυρία Ροτ Μπέρεντ και από τη Γραμματεία και ενημερωθήκαμε πάρα πολύ καλά για το έργο του ΕΜΑ που είναι πολύ παραγωγικό και το είδαμε από πρώτο χέρι. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και σήμερα, αλλά πρώτα θα δώσουμε ε, το λόγο στον Γκουίντο Ράζι για να μας κάνει την παρουσίασή του. Έχεις το λόγο Γκουίντο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους βουλευτές της Επιτροπής αυτής που μου δώσατε την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας. Η συνάντηση αυτή ακολουθεί κάποιες επισκέψεις, αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος, αντιπροσωπείας της Επιτροπής σας το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Είναι πολύ καλό για μας που ήρθατε να μας δείτε, που μείνατε μαζί μας και ελπίζω να ήταν η επίσκεψη αυτή καρποφόρα και για σας. Σήμερα, μετά από την συνάντηση αυτή, θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στην αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Γιατί προχωρήσαμε στην αναδιάρθρωση αυτή και γιατί η νέα οργάνωση ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις και στις ανησυχίες που ενδεχομένω έχετε και έχουμε εμείς. Και τέλος, θα συνεισφέρει στην ε, καλύτερη προστασία της υγείας. Στόχος μας είναι αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι ο καθένας θέλει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικός. Και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να φέρουμε σε πέρας τον ίδιο όγκο έργου με όσο γίνεται πιο λίγες δαπάνες. Όμως, ο φόρτος εργασίας μας αυξάνει συνεχώς. Αναλαμβάνουμε νέες αρμοδιότητες. Τα καθήκοντα μας αυτά δεν είναι μόνο η φαρμακοεπαγρύπνηση ή η εφαρμογή της φαρμακοεπαγρύπνησης που έτσι καλλιώς απαιτεί πολλά από μόνα της. Η δημόσια υγεία θα μας ε, απασχολήσει όλο και περισσότερο. Υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται μερικές φορές ε, στην παραγωγή Τώρα δεν χρειάζεται να το πω σε εσά τις περισσότερες φορές, τα προϊόντα αυτά μας έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν και νέα προϊόντα, αλλά και άλλα γνωστά παλιότερα. Αυτή η εξέλιξη στην ε, αλυσίδα προμήθειας είναι βέβαια μεγάλη πρόκληση για μας γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να επιθεωρούμε την είσοδο των προϊόντων αυτών, την διανομή τους και ο οργανισμός μας συνεργάζεται με διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, με τους διεθνείς μας εταίρους επίσης, προκειμένου να είναι σε θέση να φέρει σε πέρα στην αρμοδιότητα αυτή. Εάν η Ευρώπη θέλει να ελέγχει περισσότερο, ε, πρέπει να έχουμε και καλύτερη οργάνωση προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κατάρτιση, δεδομένα, ενημερωμένες πληροφορίες και να υπάρχει σύνδεση με όλα τα δίκτυα των Ευρωπαϊκών Αρχών. Νομίζω ότι σιγά σιγά προχωράμε. Έχουμε ένα τμήμα που ασχολείται με τον έλεγχο. Έχουμε 60 διαδικασίες αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να απελευθερωθούν και οι οικονομικοί αλλά και οι ανθρώπινοι πόροι. Και να μπορέσουμε έτσι να υποφεληθούμε περισσότερο. Δημιουργήθηκαν δύο μονάδες επίσης να στηρίξουν την ε, Επιτροπή ΣΕΔ για τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. και προκειμένου να καταλήξουμε σε όσο γίνεται πιο ε, βάσιμα δεδομένα και συμπεράσματα. Κάτι άλλο στο οποίο επικεντρώνεται ο οργανισμός μας έχει να κάνει με την ε, ανάγκη να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με όλους τους εταίρους, όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Νομίζω ότι πολλές από τις ε, διαδικασίες μέσα στις οποίες βρισκόμαστε έχουν να κάνουν με κάποιον εταίρο με κάποιον πυρογνώμονα, με τη βιομηχανία. Έχω την εντύπωση ότι ο οργανισμός αυτός φαρμάκων συλλέγει έτσι καλύτερα δεδομένα. Και η βάση αυτή δεδομένων πρέπει να ξέρετε ότι έχει συλλέξει στοιχεία κατά τη διάρκεια 20 ετών που χρησιμοποιούνται κατά διαφορετικές στιγμές και για διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό που σήμερα χρειάζεται, πιστεύω, είναι μια πιο γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Είναι πολύ βασικό για τους πάνω από 3.000 αντιπρόσωπους και πυρογνώμονες που χρησιμοποιούν τη βάση αυτή δεδομένων για να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Επίσης, υπάρχει η φαρμακοεπαγρύπνηση, αλλά πηγαίνουμε και πιο πέρα από εκεί. Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε να γίνει η πρόσβαση στη βάση αυτή δεδομένων πιο φιλική ακόμα για αυτούς, για την καθημερινή τους δουλειά. Επ' αυτού λοιπόν η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλη. Χρειάζεται μεγάλη επένδυση. Την κάναμε λοιπόν για να αναδιορθώσουμε ακριβώς την αρχιτεκτονική της βάσης αυτής δεδομένων μας, διατηρώντας βέβαια και την συνέχεια. Από 20.000 βάσεις δεδομένων περίπου, οργανώνουμε τα δεδομένα μας βάσει τεσσάρων ε, πυλών που έχουν να κάνουν με την ουσία, με την οργάνωση των προϊόντων, την αναφορά και πρόκειται για τη μεγαλύτερη πηγή δεδομένων στον τομέα αυτό παγκοσμίω. Έτσι μπορεί να μας χρησιμοποιήσει όποιο θέλει, να ψάξει τη βάση δεδομένων αυτών και να ψάξει να βρει αυτό που χρειάζεται. Επίσης έχουμε καθιδρύσει και μια διακυβέρνηση πληροφορικής προκειμένου να φτάσουμε στο καλύτερο επίπεδο ολοκλήρωσης των δικτύων. Έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα όπως καταλαβαίνετε, άρα πρέπει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε για να ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα συστήματα. Λειτουργικά. Ο πρώτος γύρος θα συμπληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής. Πρόκειται για τις ουσίες. Τον πυλώνα για τις ουσίες, που είναι ο πιο σημαντικός από όλους τους πυλώνες. Τώρα υπάρχουν και νέες λειτουργίες, ιδιαίτερα για την φαρμακοεπαγρύπνηση και με αυτό θα ασχοληθούμε το 2014. Έχουμε ένα νέο τμήμα για τους εταίρους μας που ασχολείται με αυτούς και ένα νέο τμήμα που αφοσιώνεται στην ενσωμάτωση των δεδομένων εσωτερικά και εξωτερικά και με τη διαχείρισή τους. Όπως σας είπα, η ασφάλεια είναι για μας μεγάλη προτεραιότητα. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το θέμα της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε για τη δημόσια υγεία και γι' αυτό θέλουμε να ασχοληθούμε με την καινοτομία. Να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τις φαρμακευτικές ανάγκες. Ξέρετε ότι η καινοτομία είναι μια περίπλοκη διαδικασία. αλλάζουν τα μοντέλα το blockbuster στο πιο προσωποποιημένο, εξατομικευμένο φάρμακο. Αλλάζουν ε, οι ενδιάμεση, τα διάφορα σώματα. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά δεδομένα να μπορούμε έτσι να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την απολυσματικότητα όταν τα προϊόντα αυτά περάσουν στην αγορά. Για να γίνει αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον το οποίο αλλάζει, άρα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Γι' αυτό και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προσπαθεί να περάσει από μια ενδιάμεση περίοδο και να καταλήξει σε ένα νέο μοντέλο σχέσεις οφέλους και κόστους, διατηρώντας βέβαια, βέβαια πάντα το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν, οι επαγγελματίες, οι ασθενείς, οι ερευνητές, οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι κλάδοι. Και αν προσπαθήσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας την καλύτερη πραγματογνωμοσύνη. Βέβαια, είναι θέμα ανταγωνισμού, έτσι πρέπει κανείς να ψάξει να βρει τους εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει μια νέα μονάδα που έχει να κάνει με την έρευνα και την ανάπτυξη. με επιστημονικά δεδομένα, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσφαση ανά πάσα στιγμή. Δίνει και τακτικά βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, ε, επιχειρήσεις και όλες τις ενότητες εκείνες οι οποίες μπορεί να έχουν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον όπου να προσφέρονται ε, επιστημονικά δεδομένα και η διαδικασία να είναι παράλληλη με εκείνη της ανάπτυξης των προϊόντων και όχι διαδοχική. Ε, μας αρέσει η ιδέα της ε, ενίας στηρίδας, προκειμένου να προσφέρουμε ε, καλύτερα και σφαιρέστερα φάρμακα, τόσο για ανθρώπινη χρήση όσο και για τα ζώα. Θα μπορούσα να συνεχίσω πάρα πολύ, αλλά προτιμώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, ό,τι ερωτήσεις έχετε, είμαι στη διάθεσή σας. Συνεπώς, θα ολοκληρώσω πάλι αναγνωρίζοντας τη βοήθειά σας, ευχαριστώντας σας για την βοήθεια και την εμπιστοσύνη που προσφέρετε στον οργανισμό μας και στο δίκτυο φαρμάκων. χρειαζόμαστε την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας στις αλλαγές αυτές που κάνουμε εγώ και συναδελφοί μου. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας, της παρούσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλλον είναι τελευταία φορά που έρχομαι εδώ. Με την Dagmar Rod Berendt βέβαια έχουμε συνεχώς επαφές. Εκείνη ήταν πάντα το σημείο επαφής για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αλλά επιπλέον μπόρεσε και μας πρόσφερε πάρα πολύ βοήθεια, στήριξη, συμβουλές, επικοδομητική κριτική, ε, μας προειδοποίησε πολλές φορές. Γενικά βοήθησε τον οργανισμό όσο δεν φαντάζεστε. Οπότε ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα στην Dagmar, δεν ξέρω αν θα είναι εδώ στο επόμενο κοινοβούλιο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής σας επίσης για τις συνεχείς προσπάθειες της και τέλος τον Ματίας Χρότε και όλους τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής αυτές, για, αυτής για την βοήθειά σας, τη στήριξή σας και την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κιντοράζη για τα καλά σας λόγια και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Έχουμε εδώ δύο εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου, τον καθηγητή Τζουζέπε Τιστίκο και τον καθηγητή Λέμαφ. Ζητούν το λόγο και οι δύο με τη σειρά που ανέφερα. Καταρχήν, Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κουίντο Ράζη και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι παρά τις δυσκολίες που βιώνουμε λόγω της οικονομικής κρίσης, η διαχείριση του οργανισμού φαρμάκων ε, γίνεται σωστά γιατί και αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των 7 ε, επιτροπών, γιατί παλιά θα θυμάστε ότι κάθε επιτροπή δούλευε μόνη της. Τώρα υπάρχει συντονισμός, υπάρχει συνέργεια μεταξύ των ε, επιτροπών που οδηγεί σε ενδιαφέροντα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω επίσης, ευχαριστώ πολύ Φρανσουάζ, η άξια μητέρα της ε, φαρμακευτικής νομοθεσίας, θα θυμάμαι αυτά. Να ευχαριστήσω λοιπόν επίσης ε, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φαρμάκων γιατί δέχτηκαν την πρότασή μου. Με άλλα λόγια, δέχτηκαν να αλλάξουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Γιατί μέχρι τώρα οι κλινικές ε, δοκιμές για το, την νόσο του Αλτσχάιμερ και αυτό είναι πρόβλημα. Πρόβλημα μεγάλης σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ασθενείς, τις οικογένειες, τον Ευρωπαίο πολίτη. Μέχρι τώρα λοιπόν δαπανίσαμε χρήμα επί μια δεκαετία, δαπανίσαμε χρόνο, χωρίς να βγουν καινούργια φάρμακα. Γιατί, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές ήταν λάθος. Δεν μπορεί να ε, δεν μπορεί να επιζητούμε να αντιστραφεί η πρόοδος της νόσου, η εξέλιξη όταν έχουν καταστραφεί εκατομμύρια νευρώνες ήδη. Αυτό δεν γίνεται. Πρότεινα λοιπόν και ο αίμα δέχτηκε να γίνονται κλινικές δοκιμές στην έναρξη της νόσου του Αλτσχάιμερ. Με άλλα λόγια, όταν πια υπάρχει, όταν, ε, υπάρχει μόνο μια ήπια γνωσιακή διαταραχή. Γιατί μόνο τότε και με τη βοήθεια των διαδικασιών του οργανισμού θα έχουμε μια γρήγορη διαδικασία, αλλιώς δεν θα τελειώσουμε. Αν κρατήσουν πολύ οι, οι, μελέτες, δεν θα ε, καταλήξουμε. Ενώ είναι οξία η ανάγκη και χρειάζονται νέες θεραπείες. Είναι σημαντικό λοιπόν να αλλάξει η διαδικασία διοδότησης και με την ταχεία διαδικασία που τη δέχεται και ο FDA, άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε στην Ευρώπη. Και ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί αυτό θα είναι το έργο του επομένου κοινοβουλίου, μπορεί και να μην είμαι, δεν ξέρει κανείς. Υπάρχει πάντως ανάγκη να ξανασυζητηθεί η σημασία της Επιτροπής για προχωρημένες θεραπείες. Μέχρι τώρα ε, είναι όδινεν όρος και έτεκεν μην δηλαδή ε, και τρώνε πολλά χρήματα Πρέπει λοιπόν να δουλέψουν διαφορετικά, να βγάζουν περισσότερο ίσως ε, υποβοηθούμενοι από μια καινούργια νομοθεσία, ώστε να έρθουν οι αρμόδιοι και να μείνουν στην Επιτροπή HAPP. Εγώ χαίρομαι που βλέπω πολλούς φίλους, ε, πραγματικά νιώθω ενθουσιασμό που σας έχουμε μαζί μας και ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και ο κύριος Λέμερ τώρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια για την συνεργασία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Ράζη και του προσωπικού του οργανισμού. Ο Γουίντο Ράζη έκανε μια εσωτερική αναδιοργάνωση της ΕΜΑ, είπε ότι χρειάζεται, είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ ένα σαφέστατο κανονισμό που θα διέπει το θέμα αυτό, τη σύγκρουση των συμφερόντων. Επιτρέψτε μου όμως δύο λόγια που μπορεί και να είναι κέρια. Εγώ είμαι από την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξετάζοντας τη σύγκρουση συμφερόντων που συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, βλέπω ότι υπάρχει επίπεδο κινδύνου δύο ήδη, αν ένας ε, οργανισμός ε, πάρει κάποια χρηματοδότηση. Ε, αυτό είναι ασαφές όμως ο ορισμός και επειδή είμαι πανεπιστημιακός και δεν ξέρω αν εδώ εννοούμε το Ινστιτούτο Φαρμακολογίας ή κάποια σχολή ή κάποιο πανεπιστήμιο, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν αδύνατον για οποιονδήποτε από την ακαδημαϊκή κοινότητα να πάει και να υπηρετεί, συνεργαστεί στον οργανισμό φαρμάκου. Αν ένας συνάδελφος σε ένα τμήμα ή σε μια σχολή παίρνει μια επιχορήγηση, τότε βρίσκεται σε επίπεδο κινδύνου 2. Αυτό είναι λοιπόν αδύνατον. Εμείς αναλαμβάνουμε ευθύνη ατομική και όχι για όλο το... όλα τα όργανα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συζητήσουμε και να το διευκρινίσουμε. Υπογραμμίζω και πάλι ότι υπογραμμίζω απόλυτα το θέμα αυτό για τη σύγκρουση συμφερόντων, αλλά το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να επαναξιολογηθεί θεωρώ. Δεύτερο σημείο, πολύ βαρύ θέμα που ασχόλησε το διοικητικό, είναι η συζήτηση των κανονισμών για τα καύσιμα και πώς θα διασφαλίσουμε την αηφορία των ε, δικτύων φαρμάκων. Εδώ χρειάζονται σαφείς ορισμοί, ε, διαχωρισμοί ευθυνών, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο ανέφερε στη συζήτηση που έκανε ότι η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ε, συζήτηση για τους κανονισμούς. Δεν θα θίξω το θέμα της ευθύνης του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα επιμερίσουμε τις ευθύνες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ρύθμισης των αμοιβών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των οργανισμών. Ευχαριστώ. Ε, όχι κανονισμός για τα καύσιμα, συγγνώμη, για τις αμοιβέ. Ε, λοιπόν, ε, εδώ δίνουμε το λόγο στους ομιλητές. Ε, τελευταία η κυρία Κουστέχα ζήτησε το λόγο. Ε, νομίζω ότι ανέφερα τα ονόματα όλων όσων ζήτησαν το λόγο. Α, η κυρία Γιανακουδάκη, δεν την ανέφερα. Η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλος πειρασμός να αναφερθώ σε πολλά πράγματα, αλλά βλέποντας ποιοι ζήτησαν το λόγο, ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα πω εγώ όλα. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Γκουίντο Ράση, όχι μόνο για τα πολύ καλά του λόγια, αλλά επίσης και για αυτά που παρουσιάσατε εδώ. Πρέπει να ομολογήσω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του ε, αίμα. Ε, πιστεύω ότι μπορεί να είστε πολύ περήφανος για αυτόν τον οργανισμό. Είναι ένας από τους καλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη, ίσως και παγκοσμίως, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονταν κάποιες αλλαγές, γιατί όπως αναφέρατε ήδη, πώς το είπατε, Τι κριτική ήταν αυτή, συμπαθητική. Α, επικοδομητική κριτική. Ναι, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπες. Λοιπόν, ίσως στο παρελθόν δεν ήταν η κριτική τόσο επικοδομητική. Η διαδικασία λοιπόν αυτή αναδιάρθρωση στον οργανισμό χρειαζόταν πραγματικά. Είναι επίσης ένα καλό μήνυμα για όλους, ένα καλό σημάδι σε μια περίοδο μικρότερων προϋπολογισμών ε, να δουν πώς μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Και θα επανέλθω σε αυτό σε δύο λεπτά, όπου ίσως θα πρέπει να διαφωνήσουμε ελαφρώς με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι ε, των ε, Εθνικών Αρχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πιστεύω ότι το μήνυμα ενός οργανισμού που αναπτύχθηκε μεταξύ και έχει μεγάλη επιρροή σε όλο τον κόσμο, είναι καλό να δείχνει ότι ο οργανισμός αυτός εξετάζει προσεκτικά τους πόρους του και πώς τους δαπανά. Πριν έρθω στο θέμα των αμοιβών, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια για τη λειτουργία συνολικά του αίμα. Είναι και ο Πέτερ εδώ που είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου για τη δουλειά. Θεωρώ ότι η αξιοπιστία του αίμα σχετίζεται ε, με τα δεδομένα που ε, παρέχει ο αίμα. Κοιτάζοντας λοιπόν ε, το σύστημα το μηχανογραφικό ε, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν παράδειγμα αποτελεσματικότητας ε, μας στο παρελθόν και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι έγινε με τα σχετικά κονδύλια πριν αναλάβετε εσείς ως ε, εκτελεστικός διευθυντής τελικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε βάση δεδομένων, όχι μόνο για τις κλινικές μελέτες, αλλά και για την φαρμακο, φαρμακοεπαγρύπνηση, θα πρέπει να λειτουργήσουν όλες αυτές οι βάσεις δεδομένων όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ αν θα μπορούσε να μας καθησυχάσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και ως προς τις κλινικές μελέτες, ίσως και ο Σούσα το επαναφέρει αυτό το θέμα, οι πολίτες, οι ε, γιατροί, οι ασθενείς όλοι έχουν ε, σαφές συμφέρον για μια καλή λειτουργία της, ε, των βάσεων δεδομένων. Τώρα για την φάρμακο ε, φάρμακοεπαγρύπνηση. Καθώς ο συνάδελφος δεν μπόρεσε να είναι εδώ παρούσα και αυτό ίσως συνδέεται εν μέρη και έμεσα με το θέμα των αμοιβών, θα μπορούσαμε να δούμε την κατάσταση των ε, επισημάνσεων για την φαρμακοεπαγρύπνηση για όλα τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να μας ε, ε πεις από τώρα κάποια σχετικά στοιχεία ή και κάποια προσωπικά σχόλια αν έχεις. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε και να λέμε και στους πολίτες μας ότι τα φάρμακα υπάρχουν για να βοηθούν και να θεραπεύουν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα 100% ασφαλές φάρμακο, όπως δεν υπάρχει κανένα 100% ασφαλές χημικό. Όλα έχουν τις ανεπιθύμητες ε, δράσεις και κάτι που φαίνεται καλό σήμερα μπορεί σε 10 χρόνια να αποδειχθεί ότι παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Ε, το ότι αναπτύσσεται η επιστήμη είναι καλό για μας όταν αποδεικνύει κάτι που δεν το ξέραμε πριν από 10 χρόνια και με χαρά μου ε, σε άκουσα να αναφέρεσαι στην καινοτομία από τη μια μεριά και στις ε, ε, ιατρικές ανάγκες από την άλλη γιατί δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές οι ιατρικές ανάγκες είναι κάτι το διαφορετικό από την καινοτομία. Και τέλος, θα ήθελα να έρθω στο θέμα της ρύθμισης των αμοιβών. Ο κύριος Λέμαν είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να έχει λόγο γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ενός οργανισμού. Θα πάρει τον προϋπολογισμό και την νομοθεσία όπως έχουν. Εσείς όμως που είστε στο νομοθετικό σώμα, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να είστε οι πρώτοι που θα έπρεπε να υποστηρίξετε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σαφής λοιπόν η απάντηση. Ναι, όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει λόγο. Θα πρέπει να πάρει τα πράγματα όπως του έρχονται. Τώρα, για το ερώτημα το κατά πόσον ένα δίκτυο ιατρικό, ρυθμιστικό, έχει μία προστιθέμενη αξία. Μπορεί αν ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Αν οι εθνικοί φορείς χρησιμοποιούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό μόνο όταν τους βολεύει, όταν είναι η σωστή περίπτωση μάλλον, και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όταν είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας, πιστεύω ότι οι, εθνικοί, οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν να κάνουν τη δουλειά τους. Το πραγματικό ερώτημα είναι, εκπληρούν τα, τα καθήκοντά τους. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα διαδικασία αδειοδότησης ή μια νέα διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης και υπάρχει ένας εισηγητής από ένα κράτος μέλος, αυτός ο εισηγητής όταν παίρνει πραγματικά σοβαρά τη δουλειά του και ε, κάνει ε, τη δουλειά του με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, πολύ ωραία. Αν όμως ο εισηγητής δεν μπορεί να το κάνει αυτό και η γραμματεία του αίμα πρέπει να κάνει την πραγματική δουλειά ή πρέπει να μεταφράσει, ε, πραγματικά τότε υπάρχει ένα κενό προφανώς. Τώρα αν στη συνέχεια το κράτος μέλος πιστεύει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει τις εθνικές του ανάγκες μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από την πίσω πόρτα, λέω όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ και θέλω οι συνάδελφοι να το καταλάβουν αυτό και εσείς παρακαλώ. Ότι από τη μια μεριά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, περικόπτει τα κονδύλια για τον αίμα όπως και για όλους τους άλλους οργανισμούς καθώς επίσης και το προσωπικό κατά 5% που όπως είναι υποχρεωτικό για το υπόλοιπο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ε, ισχύει παντού στα κράτη-μέλη εξάλλου. Και από την άλλη μεριά τα κράτη-μέλη να θέλουν να παίρνουν μέσω αμοιβών ή ε, τέτοιων κονδυλίων για εκθέσεις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τους εθνικούς εμπειρογνώμους, για τους εθνικούς οργανισμούς, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να τα δεχτούμε πρέπει να χρηματοδοτήσουν τους εθνικούς, ε, να χρηματοδοτούν τους εθνικούς τους οργανισμούς τα ίδια τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά κάτι ε, δεν πάει καλά. Δεν μπορούν με τη σύνταξη εκθέσεων και με εισηγητές κλπ. να θέλουν να καλύψουν τα κενά του προϋπολογισμού τους. Από την άλλη μεριά, ένα-δύο μικρότερα κράτη-μέλη, αλλά και μεγαλύτερα, ίσως και το δικό μου το κράτος, πιστεύουν ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να μιλούν για χρήματα και όχι για ποιότητα. Να μιλούν για, και για την ποιότητα των εθνικών αδειών, για χρήματα και όχι για τις ευθύνες τους όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και θέλω να το πω όσο πιο καθαρά γίνεται, ότι οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να παίρνουν χρήματα μόνο για δουλειά που πραγματικά κάνουν. Και στη σχετική νομοθεσία πρέπει να το καθιστούν Φτάμε απολύτω σαφές ότι οι εθνικές αρχές όταν πληρώνονται για του συζητητέ του, πρέπει να ξεκαθαρίζουν πάρα πολύ καλά τι δουλειά κάνουν. Αν αντίθετα πρέπει να πούνε ότι ο, ο αίμα πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, τότε ξεκινάμε από λάθος σημείο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε ένα κενό, ένα χάσμα εδώ, να μην υπάρξει ε, ε, ένα λάθος είδος ανταγωνισμού ανάμεσα στους εθνικούς οργανισμούς και τον αίμα που δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Και ε, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι γίνεται εδώ με την επιμέρους νομοθεσία και ακούμε και με πολύ προσοχή τα σημάδια που έρχονται από την Ολλανδία και από άλλες χώρες. Στην Αγκουτιέρες, Κορτίνες. Η ε, κυρία Κορδίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εδώ παλιού φίλου και τον καθηγητή νηστικό με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων όπω άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει όμω κάτι που με απασχολεί. Πάντα με απασχολεί εδώ. Σε τι βαθμό η νομοθεσία την οποία αποφασίζουμε εδώ μπορεί να εφαρμοστεί. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζεται η νομοθεσία. Οπότε, με την φαρμακοεπαγρύπνηση πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μήπως είναι υπερβολικά περίπλοκα και δεν εφαρμόζονται. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστούμε. Μαργαρίτα Ούκεν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Κύριε Ρώση, ευχαριστώ και για την παρουσία σας. Δύο σχόλια έχω. Πρώτον, το ένα είναι αυτό που είπε ο κύριος Λέμα για την σύγκρουση συμφερόντων. Είμαστε ιστερικοί πια με το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Πάρα πολλά χρήματα κυκλοφορούν και έχουμε δει τι γίνεται είναι θέμα εμπιστοσύνη των πολιτών. Χάνουμε την αξιοπιστία μας. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για φάρμακα δεν βρίσκονται μέσα σε καμία σύγκρουση συμφερόντων. Να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Αυτά έχουμε ζητήσει. Στην Επιτροπή Αναφορών, που είμαι μέλος, πολλές φορές συζητάμε για νέα ρύθμιση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων που θα καλύπτει και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων με ρύθμιση όσον αφορά την χρηστή διαχείριση και εκεί περιλαμβάνεται και το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Στη Δανία έχουμε κάποιες κακές εμπειρίες, μία είναι πολύ κακή. Στην Ελλάδα για τα ε, γενώσιμα φάρμακα η Ελλάδα που υποφέρει τόσο πολύ από την οικονομική κρίση και με διαφθορά, όπως θέλετε πείτε το, αν υπάρχει θέμα συμφέροντος με κάποιον πρέπει να είναι μακριά από εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. τι εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούμε. Όντω, να μην είναι εμπλεγμένοι με τη βιομηχανία. Αυτό πρέπει να το διασφαλίζουμε. Έπειτα για τη διαφάνεια, τουλάχιστον στον τύπο της Δανίας, που ξέρω ότι είσαστε εδώ σήμερα, έχουν ήδη ασχοληθεί και ρωτάνε, με πήραν και τηλέφωνο, αν υπάρχουν νέα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που εισάγατε μετά την υπόθεση που είχαμε με τον Ombudsman, όπου το Northern Institute έγινε αναφορά δηλαδή στον Ombudsman, όπου έλεγε ότι το θέμα της διαφάνειας πρέπει να ευνοεί τον ασθενή και όχι την βιομηχανία. Και ο Ombudsman έδωσε συνέχεια στην αναφορά αυτή και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, αλλά μετά στο δικαστήριο κόλλησε. Παρακάνθηκε ο Ομπουτσμαν όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες κτλ. Όλα αυτά πήγαν περίπατο. Λοιπόν, θα ήθελα να έχω κάποιες απαντήσεις να πάω στη χώρα μου όταν γυρίσω. Πόσο καιρό ακόμα θα αναβάλλετε. Το θέμα αυτό των ασθενών, του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας, πόσο καιρό ακόμα θα καθυστερεί και δεν θα είναι πάνω από τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Υπάρχουν φάρμακα που έχουν άδειες, έχουν τα πάντα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια πρέπει να επιμείνουμε. Και ελπίζω ότι μπορείτε να μου δώσετε κάποιες απαντήσεις, να μου πείτε ότι έχουμε προχωρήσει και ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλα δύο-τρία χρόνια. Έχουμε τους δύο-τρεις κανονισμούς εδώ στο Κοινοβούλιο για τις δοκιμές, τα φαρμακευτικά μηχανήματα κλπ. Θα είναι μεγάλη πρόοδος για όλο τον κόσμο και για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρώπη, αν προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε, Μαργαρή Τόκεν. Η κυρία ε, Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να πω ευχαριστώ στον κύριο Ρώση για την παρουσία του εδώ, για όσα μας είπε όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της δουλειάς του και την αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η δικιά μου πολιτική ομάδα και εγώ ίδια που είμαι από την ομάδα της ΓΚΟΕ και ε, Βόρεια Αριστερά είμαστε κατά της ιδέας περικοπής 5% στις διοικητικές δαπάνες. θέλουμε μια πιο φιλόδοξη εμείς πρόταση για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζαμε λοιπόν σε ένα προπολογισμό πιο φιλόδοξο και για την επόμενη χρονιά το 2014 αλλά και για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Συνεπώς, δεν είμαι σύμφωνη με τις περικοπές αυτές και το εκδηλώνω αυτό και με την ψήφο μου. Στην Πορτογαλία συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει θαύματα με το τίποτα. 5% περικοπή από πού θα κόψουμε. Λέτε από τους πόρους. Ναι, αλλά όχι και από τις αρμοδιότητες. Οπότε πώς θα γίνει αυτό. Αυτό που μου άρεσε πολύ που είπατε είναι η τράπεζα δεδομένων. Πιστεύω ότι είναι κάτι ουσιώδες, θεμελιώδες και η βελτίωση αυτή που αναφέρατε όσον αφορά τη σύνθεση και τη δομή της τράπεζας δεδομένων είναι το πιο σημαντικό. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει μια τράπεζα δεδομένων για τους πολίτες είτε είναι ήδη ασθενείς είτε δεν είναι, και για όλους τους επαγγελματίε της υγεία, για όλους τους ερευνητέ επίσης. Γι' αυτό λοιπόν οι βελτιώσει αυτές που επιφέρετε και η προσπάθεια αυτή που μα είπατε ότι κάνετε για να είναι πιο εύκολη πρόσβαση στην τράπεζα αυτή δεδομένων, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε συγχαρητήρια γι' αυτό. Αλλά μην ξεχνάτε την ερώτησή μου. Από πού θα κόψετε, πώς θα κάνετε αυτές τις περικοπές. Αυτό θέλω να πείτε. Αφού σα υποχρεώνουν να κόψετε από πού. Γιατί τέτοιε περικοπές έχουν άμεσε επιπτώσεις. Το είπε και η κυρία Όκεν ότι η διαφάνεια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η διαφάνεια των δεδομένων, των μελετών, των αποτελεσμάτων. Εντάξει, δεν θέλω να γκρινιάζω υπερβολικά, αλλά έχω να σας κάνω και δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να ακούσω την άποψή σας. Τους τελευταίους μήνες εδώ στην Επιτροπή αυτή ασχολήθηκα με τρία σημαντικά πιστεύω θέματα. Νομοθετικά έχουν μεγάλη σημασία οι κλινικές ε, δοκιμές, τα υγειονομικά προϊόντα και in vitro δοκιμές. Όλα αυτά τα θέματα είναι ζωτική σημασίας για να διασφαλίζουμε την προστασία των ε, ασθενών. Άρα χρειαζόμαστε ε, γερές έρευνες για να προσφέρουμε διάγνωση ποιότητας. Οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια ήταν ικανοποιητικές όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές και τα γενομικά προϊόντα. Η πρόταση που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή αυτή την Τετάρτη ήταν καλύτερη από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραμένουν όμως κάποιες αδυναμίες δεν είναι σαφής η θέση όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές. Η ανάγκη δηλαδή να υπάρχει έγκριση και όχι μόνο εξέταση ή ανάλυση ενός πρωτοκόλου κλινικής δοκιμής από την Επιτροπή Ηθικής. Πρέπει να γίνεται η ανάλυση πριν ξεκινήσει η δοκιμή αυτή. Πρέπει να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή αυτή πριν περάσουμε στην εφαρμογή. Γι' αυτό και έρχομαι στις δύο συγκεκριμένες μου ερωτήσεις. Πρώτον, για τα υγειονομικά προϊόντα. Ποια είναι η γνώμη σας. Υψηλού κινδύνου, ε. Ποια είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε εμείς για να διασφαλίσουμε υψηλό βαθμό προστασίας στους ασθενείς μας στην Ευρώπη. Πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου ποιος είναι ο καλύτερος μηχανισμός για να διασφαλίσουμε την προστασία αυτή των ασθενών. Δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικά με τις κλινικές δοκιμές. Πριν από λίγα χρόνια η Τράπεζα Δεδομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων μάλλον μετά από λίγα χρόνια θα μπορεί να περιλαμβάνει ε, δεδομένα που δεν θα έχουν περάσει από την Επιτροπή Ηθικής. Και αυτή είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση και θέλω να έχω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω στον κύριο Ράση ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να ακούσω την παρουσίασή του στην αρχή γιατί ήμουνα όχι μακριά από εδώ αλλά δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Λυπάμαι γι' αυτό. Πάντως θέλω να του πω επίσης ότι έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου ότι είχα την ευκαιρία όπως και άλλοι συνάδελφοι να συμμετάσχω σε επισκέψεις που κάναμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και να συμμετάσχω εκεί σε συνεδριάσεις και θαύμασα κάθε φορά τα όσα μάθαμε και είδαμε εκεί. Θέλω να σας πω ότι το έργο σας το βρίσκω πολύ σπουδαίο και ότι εξεπλάγει από την υψηλή ποιότητα των εργασιών σας. Λοιπόν, και εγώ λυπάμαι για τη μείωση αυτή στον προπολογισμό κατά 5%. Δεδομένου μάλιστα ότι σας ζητούμε όλο και περισσότερα. Σας ζητάμε να κάνετε περισσότερα πράγματα, περισσότερη δουλειά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχεια απευθύνεται σε εσά και σας αναθέτει όλο και περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Οπότε η μείωση αυτή στον προπολογισμό δεν σας επιτρέπει να τα αποκριθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεπώς είσαστε υποχρεωμένοι αναγκαστικά να ε, ζητήσετε αμοιβή. Και εκεί είναι που ερχόμαστε στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι λοιπόν μια κατάσταση περίπλοκη. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει μια καλή διέξοδο. Και ανησυχώ γιατί εντάξει σύγκρουση συμφερόντων τελικά τη βρίσκουμε λίγο πολύ παντού. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση εργασίας. Αλλιώς είναι αδύνατον να κάνετε τη δουλειά σας. Και κινδυνεύετε επίσης να χάσετε ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία και πραγματογνωμοσύνη επειδή υπάρχει κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων. Εντάξει, εγώ θέλω να υπάρχει διαφάνεια, φυσικά, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να μην σας εμποδίζει η προσπάθεια αυτή να κάνετε σωστά τη δουλειά σας και να έχετε στη διάθεσή σας τους εμπειρογνώμονες που χρειάζεται. Οπότε με κάθε ειλικρίνεια θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε από αυτού. Θέλω να μας πείτε, τελικά πιστεύετε ότι πάμε πάρα πολύ μακριά στο θέμα αυτό της σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει τη δυνατότητά σας για να φέρετε σε πέρα στα καθήκοντά σας. Χαίρομαι που έχουμε εδώ και τους εκπροσώπους, ιδιαίτερα τον καθηγητή που ήταν και συνάδελφος ε, εδώ, λαμπρός συνάδελφος για αρκετά χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε ότι παρακολουθεί και εκείνο ε, το έργο σας. Λοιπόν, όσον αφορά τις αμοιβέ αυτές που πληρώνονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, με αυτή τη χρηματοδότηση, πείτε μας τη γνώμη σας. Αυτοί που έχουν την άδεια διάθεση στην αγορά, μήπως τελικά πληρώνουν δύο φορές παραπάνω είτε στα κράτη-μέλη είτε στον οργανισμό για την ίδια δουλειά, για την φαρμακοεπαγρύπνηση, μήπως υπάρχει επικάλυψη εκεί, εδώ υπάρχει κάποιο λάθος ή όχι. Κάθε είσοδος στην βάση δεδομένων ε, πληρώνει τέλη. Σωστά. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού Πιστεύετε ότι έχει κάποια όρια? Γιατί μπορεί να υπάρξουν πολλέ είσοδοι που έχουν να κάνουν με το ίδιο φάρμακο, γιατί μπορεί να θέλει κανεί να δει τη συσκευασία, τη δόση κτλ. Οπότε αυτό που ε, μπαίνει στη βάση δεδομένων πρέπει να πληρώσει πολλέ φορέ τα τέλη αυτά. Και κάτι που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Και εγώ το είπα όταν είχα έρθει να σας δω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ολομέλεια τη 2η του Οκτωβρίου υιοθέτησε ένα κείμενο για την προστασία των ασθενών με την οποία ζητάει κατευθυντήριες γραμμές από τον οργανισμό για τη χρήση των φαρμάκων. Λοιπόν, θέλω να ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό. Τι σκοπεύετε να κάνετε, μια που υπήρξαν ε? διάφορες περιπτώσεις με το Μεδιατόρ στην Γαλλία ή άλλο φάρμακο στη Δανία. Οπότε θέλω να ξέρω εσείς πώς θα πλαισιώσετε την χρήση αυτή των φαρμάκων που βρίσκονται εκτός. Αμέν. Η κυρία Κουδάκη τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Που με ξεχάσατε όμως. Εγώ είχα έρθει και στην επίσκεψη και μου άρεσε πολύ και έμαθα και πολλά. Γυρίζω στην ε, δήλωση ότι δεν κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Το λέμε εμείς. Ε, ε, βέβαια χρειάζεται για να κάνεις ομελέτα να αγοράσεις και αυγά πριν να τα σπάσεις. Και μερικοί συνάδελφοι έχουν πρόβλημα αγορών. Πήγα στην Ελλάδα πρόσφατα, Έχουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, να τα ξέρουμε αυτά. Εδώ μιλάμε για λεφτά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, έχουν, πήγα σε ένα φαρμακείο στην Ελλάδα το περασμένο Σαββατοκύριακο, έχουν κάποια γενώσιμα. Τέλος πάντων, εγώ σας συνεχάριν για το 5% και προσβλέπω παρόμοιες περικοπές στο μέλλον, ενώ θα περνάμε από αυτή την ζώρικη περίοδο για όλη την Ευρώπη επικοδομητική η κριτική μου. Τώρα, ή τα τέλη φαρμακοεπαγρύπνησης ε, με έχουν απασχολήσει και υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Καταρχήν ο οργανισμός σας παίζει μεγάλο ρόλο εδώ. Γιατί ε, ε, φροντίζει για έναν έλεγχο με τις αρμόδιες αρχές και έχετε και ένα σύστημα μηχανοργάνωσης που θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν έχει στηθεί όμως ακόμα και μπορεί να καθυστερήσει, οπότε θέλω να σας ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό. Επίσης χάρηκα πολύ διότι ε, τα τέλη που πρότεινε η Κομισιόν ε, λέτε ότι δεν χρειάζονται, μπορεί να κάνετε τη δουλειά και με λιγότερα. Θαυμάσια. Ε, ε, ε ελπίζω να τα ε, τηρήσετε όλα αυτά, γιατί καμιά φορά είναι δύσκολο. Ελπίζω να κρατήσουμε το μικρότερο ποσό. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση, αν θα μείνουμε στο μικρότερο ποσό και αν είναι έτοιμο το σύστημα μηχανοργάνωσης. Ευχαριστώ. Εγώ ποτέ δεν θα σας, θα σας ξεχνούσα και ούτως ή άλλως ποτέ από τη λίστα των αγοριτών. Ο Γκουίντο Ράζι τώρα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις, να σχολιάσει τις προτάσεις κλπ. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, το καλύτερό μου, για να τα απαντήσω όλα. Αν ξεχάσω τίποτα, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά να μου το επισημάνετε αυτό. Λοιπόν, με τη σειρά Ορισμένες ε, θα τις ομοδοποιήσω γιατί είναι παρόμοιες οι ερωτήσεις. Ο κύριος ε, ο καθηγητής Λέμερ ε, είπε δύο πράγματα ουσιαστικά. Το ένα αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων του εμπειρογνώμονα και αυτό το θέμα το έθεσαν και πολλοί άλλοι. η κυρία Ροτ Μπέρεντ, η κυρία Άουκεν, η κυρία Σόουσα και η κυρία Γκροστέτ. Λοιπόν, ποια είναι τα τελευταία νέα. Ε, εμείς στη συνάντηση με αυτό το θέμα έπρεπε να έχουμε ε, μια ισορροπία μεταξύ των καλύτερων εμπειρογνωμόνων που θα έπρεπε να έχουμε και ταυτόχρονα να αποδώσουμε σημασία και στο άλλο θέμα να μην υπάρχουν παρεμπολές που θα επηρεάσουν την αξιοπιστία του συστήματος και την εμπιστοσύνη σε αυτό. Να συνοψίσω την προσωπική μου άποψη και το συμπέρασμα της συνάντησης όπου μας απασχόλησαν όλα αυτά. Ξέρουμε ότι για την ακαδημαϊκή κοινότητα χρειάζεται μια μεθοδολογία ώστε πολύ συγκεκριμένα να εντοπίσουμε κάποιο συμφέρον. Πάνω από το, τα επίπεδα κινδύνου 1 με 3 πρέπει να προσδιορίσουμε πού βρίσκεται το συμφέρον και ενδεχομένως να προλάβουμε να υπάρχει αυτό το συμφέρον. Η μεθοδολογία δεν έχει διευκρινιστεί, ακόμα την επεξεργαζόμαστε και το Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφανθεί οριστικά. Αν μειώσουμε το επίπεδο προσοχής μας, το, η σύγκρουση συμφέροντος μπορεί να ε, επικρατήσει και να αμφισβητηθεί μια απόφαση. Πρέπει να υπάρχει μια ε, ισορροπία για το χρονικό ορίζοντα δύο, τρία, τέσσερα χρόνια δεν ε, είναι ο χρονικό, το, το κατάλληλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι τελείωσε η σύγκρουση συμφέροντος πρέπει να το προσδιορίσουμε. Έξι-έξι μήνες έχει τελειώσει. θα ληφθεί μια απόφαση και θα σας δώσουμε τα στοιχεία της απόφασης μόλις τη λάβουμε στο διοικητικό για τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ε, κάνουμε δημοσιεύσεις, κοινοποιούμε στοιχεία, ούτως ώστε και εκτός του οργανισμού μας ε, κάποιοι να μας ε, επισημάνουν κάτι που δεν το έχουμε εμείς ανακαλύψει. Γιατί εμείς δεν κάνουμε αστυνόμευση, δεν είναι, αυτό ξεπερνά τη δουλειά μας και το έργο μας. Για τη διαφάνεια ε, ήδη ε, φροντίζομαι, αυξάνομαι το επίπεδο διαφάνειας, δημοσιεύομαι ημερήσια διάταξη πρακτικά όλων των ε, επιτροπών και στο τέλος του έτους θα μπορούμε να δημοσιεύουμε και τα πρακτικά από τη CHMP που δεν το κάναμε παλιά. τώρα, γιατί αν πάει στο δικαστήριο θα δούμε πώς θα αποφανθεί το δικαστήριο. Δηλαδή θα πρέπει αφενός να σεβόμεθα τις αποφάσεις και να σεβόμεθα και τις προσδοκίες που υπάρχουν ε, και να σεβόμεθα και τον νόμπουτσμαν, τον ε, διαμεσολαβητή. Ήδη κοινοποιούμε ε, έγγραφα πολλά και αυτό βέβαια ισχύει οριζόντια ως μέσον μέτρων για την προστασία της υγείας. Η προσωπική μου άποψη είναι να έχουμε μία ε, διαχείριση στην προσέγγιση αυτή της ε, ε, δημοσίευσης δεδομένων. Δεν θα γίνει αυτός σκοπός, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να δημοσιεύονται τα έγγραφα επί των οποίων αποφασίζουμε. Ε, γιατί εκεί θα πρέπει να αιτιολογούμε γιατί ελάβαμε για το συγκεκριμένο θέμα απόφαση και όταν ληφθεί η απόφαση τότε τελειώνει το θέμα. Ε, αυτά τα ε, δεδομένα γιατί να τα κρύψουμε. Μακροπρόθεσμα, ωφέλη θα έχουμε και για την ανάπτυξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Περισσότερο από τις μεγάλες εκτός Ευρώπης. Πάντως εμείς τώρα είμαστε σε στάση αναμονής. Πρέπει να δούμε τι θα πει το δικαστήριο, πώς θα αποφανθεί. Ελπίζω έτσι να κάλυψα το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων Η κυρία Ροσμπέραντ ρώτησε για το χρονοδιάγραμμα. Κατά κάποιο τρόπο... Α, για το πότε θα, επίσης θα στηθεί το σύστημα της μηχανοργάνωσης. Και η κυρία Γιανακουδάκη το ρώτησε αυτό. Είναι λίγο η ερώτηση της κότας και του αυγού. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε καλή βάση δεδομένων αν δεν έχουμε τα τέλη και πώς μπορούμε να εισπράττουμε τα τέλη αν δεν έχουμε βάση δεδομένων, αξιόπιστη. Γι' αυτό άρχισα να μιλάω λέγοντας ότι αυτή είναι μια μεγάλη επένδυση που θαραλέα αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα κάνουμε περικοπές ούτω ώστε να βρούμε τα λεφτά για να εξασφαλίσουμε την τεχνολογία που θα χρειαζόμαστε στο μέλλον. Και πού βρισκόμαστε τώρα. Όπως σας είπα, στο τέλος του χρόνου θα έχουν ξεκαθαριστεί όλες οι ουσίες. Δηλαδή από τις 18 βάσεις δεδομένων που γιατί φορτώθηκαν περίπου μισό εκατομμύριο κωδικοί με πολλές εφαρμογές, όχι πολλές αλλά πολλές τέλο πάντων εφαρμογές και κάποια σφάλματα επίσης. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα τα καθαρίσουμε όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι προσλάβαμε εξωτερικούς ε, ειδικού ε, επαγγελματίες να τα καθαρίσουν όλα αυτά, ώστε να είναι εύχριστα και να συμφωνούν και με τις λειτουργικές μας δυνατότητες για να υπάρχει δυνατότητα φάρμακο επαγρύπνησης και το δεύτερο μισό του 2014 να είναι έτοιμες οι προϋποθέσεις που θα θέσουμε και στη φαρμακοβιομηχανία. Να έχουμε προβλέψει δηλαδή τις εξελίξεις. Αυτή η εκτίμηση είναι αρκετά συντηρητική, όχι αισιόδοξη και νομίζω ότι στα μέσα του επομένου έτους θα έχουμε φτάσει εκεί. Και πολλά ακόμα θα έχουν γίνει η αλυσίδα εφοδιασμού θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Θα ήθελα η βάση δεδομένων να είναι σε λεπτομέρεια συσκευασίας και μεγέθους συσκευασίας, ούτως ώστε να προληφθούν πολλά σφάλματα γύρω από αυτό το θέμα και για τα παλιά φάρμακα. Τώρα ε, ε, κάνω μια μετάβαση για να περάσω σε ένα άλλο ερώτημα της κυρίας Ροτ Μπέρεντ. Νομίζω ότι οι παραπομπές και η νέα φαρμακοεπαγρύπνηση, όπως είπατε, τώρα προσελκύουν πολύ προσοχή. Υπάρχει αύξηση 60% των ε, σημάτων πέρσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την παραπομπή παλιού προϊόντος. Σίγουρα θα εντοπίσουμε κάτι που δεν είχε γίνει κατανοητό παλιά, αλλά μαθαίνουμε επίσης τώρα ότι πολλά προβλήματα μπορεί να προέρχονται ε, από κατασκευαστές που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα στην Ευρώπη και επίσης γίνονται και φαρμακευτικά σφάρματα και την συνταγογράφηση και όλα αυτά εντοπίζονται με την φαρμακοεπαγρύπνηση. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό των ε, ε, σημάτων που ήρθαν από κακή χρήση κάποιου φαρμάκου ε, εκτός από το φάρμακο το ίδιο. Ανοίγει λοιπόν καινούργια εποχή για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και θα μπορούμε ενδεχομένως να κάνουμε διάφορες διακρίσεις και διαφοροποιήσεις και θα μπορούμε να εντοπίζουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα του φαρμάκου, το πρόβλημα στη χρήση του και ξέροντας ότι θα ε, γίνεται η χρήση πιο περίπλοκη γιατί οι ασθενείς θα μπορεί να παίρνουν έναν ε, άπειρο συνδυασμό φαρμάκων. αυτά για τα νέα φάρμακα και που θα οδηγηθούμε με αυτά. Θα ανακαλύπτονται πιο γρήγορα. Θα μπορούμε όμως και προβλήματα να τα αντιμετωπίζουμε πολύ πιο γρήγορα. Ε, θα, για τα παλιά φάρμακα θα ε, εξειδικεύσουμε την χρήση τους ώστε να έχουμε ωφέλη και όχι προβλήματα. Επίσης η χρήση off-label που είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα. Η χρήση off-label θα καλύπτεται εν μέρη από τη νέα φαρμακοεπαγρύπνηση που θα μας επιτρέπει να ε, λέμε αν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα από την χρήση off-label και να προλαμβάνουμε αυτά που δεν θέλουμε να ε, συμβούν με τη χρήση φαρμάκων off-label. Τώρα για, το, ε, για τις, ε, τα τέλη δεν θα αποφασίσει το διοικητικό. Εσείς κυρία Ροτ Μπέρεντ είπατε, ε, μιλήσατε για τους εθνικούς αντιπροσώπους που έχουν προστιθέμενη αξία, συμφωνώ και εγώ. Θα πρέπει να διευρυνθεί η δυνατότητα του Εθνικού Φορέα να δημιουργήσει ικανότητα για ε, παγκόσμιες ε, επιθεωρήσεις ε, πρέπει να συνεργαζόμεθα οπωσδήποτε με τις τοπικές αρχές για να εξασφαλίζουμε έλεγχο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι θέλουμε να, να κάνουν εκπαίδευση ούτω ώστε να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους εκεί που χρειάζεται. Όλους τους χρειαζόμαστε και ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ικανοί, δραστήριοι, αφοσιωμένοι και πρέπει να τους αξιοποιήσουμε τώρα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η κυρία Κορτίνες μ, ρώτησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Η εμπειρία του πρώτου έτους είναι πολύ θετική και καλή. Εγώ είμαι περήφανος για τους συνεργάτες μου στον οργανισμό φαρμάκου που χωρίς ε, νέες προσλήψεις μπόρεσαν να λειτουργήσουν άριστα επί ένα χρόνο. Βεβαίως έγιναν αποσπάσεις, μεταθέσεις, ε, Οι υπερορίες βέβαια αυξήθηκαν πάρα πολύ δραστικά, αλλά είμαι πολύ περήφανος για το επίτευγμα των συνεργατών μου. Και είμαι περήφανος και για τους αντιπροσώπους και το δίκτυο, γιατί χωρίς τέλη μπορέσαμε να καλύψουμε το κόστος. Δεν μπορέσαμε βέβαια να πληρώσουμε τους εισηγητές. Και αυτό έγινε ως των επιβάσεως εθελοντικής. Και ένας μικρός αριθμός χωρών ανέλαβε ένα μεγάλο φορτίο και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κατάφερε το δίκτυο. Τώρα, πόσο θα συμπορέσουμε να το συνεχίσουμε αυτό δεν το ξέρω, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσουμε ε, στα όρια μας. Δεν μπορεί να λειτουργούμε συνεχώς ε, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Πάντως μέχρι τώρα τα κατάφερε το σύστημα. κυρία Άουκεν μου φαίνεται ότι τα είπα αυτά που ρωτήσατε για την διαφάνεια. Συγγνώμη αν ξέχασα κάτι. Ε, κυρία Σόουσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση που δείχνετε. Και δεν συμφωνείτε με το 5%. Θυμίζω όμως ότι κατά 85% στηριζόμεθα ε, από τη δουλειά, στη δουλειά μας, δηλαδή αυτοχρηματοδοτούμεθα. Δεν βαραίνουμε εμείς ε, το φορολογούμενο, σας το θυμίζω αυτό. Και γι' αυτό έχουμε 1% περικοπή, γιατί μόνο το 15% προέρχεται από ε, δημόσια κονδύλια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κάνουμε μεταθέσεις, μέχρι τώρα τα καταφέρναμε γιατί από τις 60 διαδικασίες που προανέφερα μπορέσαμε να συγκεντροποιήσουμε ήδη κάποιες για να αποφύγουμε επικαλύψεις και κάναμε ανακατανομές και νέους επιμερισμούς πόρων και έτσι επιβιώσαμε μετά την περικοπή αλλά όπως σας είπα ε, ε, δεν θα κρατήσει και πολύ αυτή η κατάσταση αν δεν βελτιωθεί το θέμα ε, ο συντονισμός επιθεωρήσεων, το η σύγκρουση συμφερόντων μας απασχόλησε γύρω στους 25 υπαλλήλους. Όλα μετράνε λοιπόν. Πάντως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών σας. Τώρα για τις κλινικές δοκιμές, τις κλινικές μελέτες, ξέρουμε ότι το θέμα συζητείται υπάρχουν και εμείς συνεπιστρόποι για αν δεν υπάρχουν ας Αυτό είναι πιθανό κίνδυνος και ε, διαρριγνύει το σύστημα συλλογή δεδομένων. Εμείς τώρα με την, τον οργανισμό μας είμαστε σε καλύτερη θέση και μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις νέες κλινικές μελέτες χωρίς πρόσθετες δαπάνες. Αυτό σημαίνει και σας διαβεβαιώνω γιατί και τώρα μας υποστηρίζει και η Κομισιόν, γιατί κάποια κράτη-μέλη ανησυχούσαν. Τέλο πάντων μπορώ να σας πω ότι ε, είχαμε δει πολλές δαπάνες να προκύπτουν από τα διαφορετικά σημεία αποθήκευσης των δεδομένων που μετά έπρεπε να μπουν στη βάση δεδομένων μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια μικρότερη επένδυση ε, η οποία θα εξασφαλίζει τη συνέπεια ευθύς εξ αρχής. Για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ να λάβουμε αποφάσεις. Πάντως, εγώ θα ήθελα πολύ να έχουμε πρόσβαση σε πραγματογνωμοσύνη, που δεν την έχουμε τώρα, γιατί υπάρχουν νέες τεχνολογίες, συστήματα ε, χορήγησης φαρμάκων, πολλά βοηθήματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι πολύ ευαίσθητα και δύσκολα στη χρήση τους ε, και χρησιμοποιούνται όμως για να χορηγηθούν τα φάρμακα. Εδώ χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη που δεν την έχουμε. Και αυτοί που αξιολογούν αυτά τα βοηθήματα πρέπει να έχουν πραγματογνωμοσύνη για τα ε, ιατροφαρμακευτικά θέματα. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Οπότε, όποια και να είναι η απόφαση, καλό θα ήταν να έχουμε μια επιτροπή όπου θα συνεδριάζουν οι εμπειρογνώμονες για να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις υπέρ της δημόσιας υγείας. Διαγνωστική in vitro. Ε, για όσους είναι συνδεδεμένοι με το Companion Diagnostics όπως λέγεται. Για αυτούς θέλουμε να έχουμε λόγο, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η ιατρική να στηρίζεται σε διάγνωση που την αγνοούμε εμείς και που δεν έχουμε καμία δυνατότητα να την ελέγχουμε. Θέλουμε να έχουμε τον τελευταίο λόγο. Εδώ, ναι, το λέω ξεκομμένα και όμα. Θέλουμε να έχουμε τον τελευταίο λόγο, ούτως ώστε να υπάρχει συνέπεια στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για τη θέση σε κυκλοφορία κάποιων ουσιών, δραστικών ουσιών. Μου φαίνεται τα απάντησα όλα, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν ξέχασα κάτι και μπορώ βέβαια να συμπληρώσω τις απαντήσεις μου και γραπτός. Ευχαριστώ πολύ Γκουιντοράζη. Νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις απαντήθηκαν. Έχουμε καλή εποπτεία τώρα του θέματος. Δηλαδή ποιο είναι το θέμα του, τι συζητείτε τώρα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, τον ΕΜΑ. Και ευχαριστώ πολύ για τη λεπτομερή παρουσίαση για τις εξοικονομήσεις, τις περικοπές, α, ως ένα βαθμό μπορεί να γίνονται. Πρέπει όμως πάντα να ξέρουμε τι κατάφερε να κάνει ο οργανισμός, γιατί του αναθέσαμε πολλά καθήκοντα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει και περισσότερα χρήματα στον οργανισμό αφού του μεταφέρει αρμοδιότητες. Διότι αν πάρει ο οργανισμός περισσότερες ε, ε, αρμοδιότητες, θα μειωθεί και η γραφειοκρατία. Δηλαδή θα μειωθεί αυξηθούν οι εργασίες των εθνικών φορέων σε τον 28. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί και χρηματοδοτικά. Δεν θα πω άλλα. Πάντως νομίζω ότι ο οργανισμός έφτασε πια στα όρια του σε ό,τι αφορά τις ε, περικοπές. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσά και τους συνεργάτες σας που ήρθαν και σήμερα εδώ ε, χαίρομαι για την καλή επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια ε, ωφεληθήκαμε πολύ από αυτό το καθεστώς. Ε, άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Jetzt möchte ich να καλωσορίσω με την ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο από το Υπουργείο Ενέργειας και Προστασίας του Κλίματος. Χαίρομαι που ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και το σημείο 6. Και εδώ πρόκειται για το νησιωτικό σύμπλεγμα Μαγιότ και το καθεστώς του. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό, όχι, λάθος, τα παίρνω πίσω όλα. Πάμε στο σημείο 5 και το Chris Davis, έκθεση εφαρμογής της, του CCS, τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα. Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την ευκαιρία που μου δίνει να συζητήσουμε κάποιες από τις ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν για την ε, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Θα θυμάστε ότι ο, Διεθνής, ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας λέει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο χρειαζόμαστε το CCS να καλύψουμε το 20% τουλάχιστον των παγκόσμιων εκπομπών, διότι διαφορετικά θα φτάσουμε σε απαράδεκτο επίπεδο θέρμανσης του πλανήτη το 2050. Η Κομισιόν λέει ότι χρειαζόμαστε το CCS αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο του 95% με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Αλλά με αυτά που κάνουν τώρα η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, ε, όπου αναπτύσσονται οι τεχνολογίες CCS, ε, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια έλλειψη ενός επιχειρηματικού μοντέλου ε, στην Ευρώπη. Και κάποιες προσδοκίες ε, υπερβολικές για το τι θα έκανε ο ιδιωτικό ε, τομέας ε, μας δείχνουν ότι θα πρέπει ή να δοθεί χρηματοδοτική βοήθεια ή να γίνουν κάποιες ρυθμιστικές απαιτήσει. Διότι το σύστημα του CCS δεν βασιζόταν ποτέ σε επιδοτήσεις όπως για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, αλλά βασιζόταν στην τιμή του άνθρακα. Υποθέτουμε ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα επένδυαν μεγάλα ποσά για να αποφύγουν τον κίνδυνο να αγοράσουν δικαιώματα εκπομπή διοξείδου του άνθρακα. Αλλά βέβαια το κόστο του άνθρακα είναι ε, αμεληταίο, άρα όλο το επιχειρηματικό μοντέλο αυτό κατέρευσε. Επίση, όταν συμφωνήσαμε για την ρυθμιστική νομοθεσία, και εγώ είμαι εξίσου υπεύθυνο γι' αυτό, όπω και οποιοδήποτε άλλο, γιατί ήμουν ο εισηγητή, επιβάλλαμε μη ρεαλιστικέ ε, προσδοκίε εκείνη την εποχή. Αν πάρουμε μια χημική βιομηχανία στην Γερμανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν πολλέ χημικέ βιομηχανίε στην ε, ε, Γερμανία που ε, εκπέμπουν παρευθείαν στην ατμόσφαιρα ε, διοξείδιο του άνθρακα. Θεωρώ ότι εσείς και η Γερμανία είστε <laughs> ένα και το αυτό. αν η Άγγελα Μέρκελ είναι η μητέρα, εσείς είστε ο θείος ή ο ξάδερφος της Γερμανίας. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο τεχνικό μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, να το δεσμεύσουμε και να το θάψουμε δύο χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης, να το εχίσουμε μέσα σε πέτρωμα, όπως κρατούσαν τα πετρώματα αυτό το μεθάνιο επιχιλιατής που το καίμε τώρα, σαν καύσιμο. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε μια χημική βιομηχανία να μην πάει απλώς σε έναν μηχανικό και να ε, του πει φτιάξε μου ένα, ε, μια κατάσταση δέσμευσης, αλλά να εγκαταστήσει και έναν αγωγό που θα φτάνει στη Βόρεια Θάλασσα και θα αναλάβει την έχηση αυτή μέσα στο πέτρωμα. Αυτά τα κάνουν ε, οι εταιρείε φυσικού αερίου, όχι οι χημικές βιομηχανίες. Είναι ένα διαφορετικός κλάδος. Άρα θα πρέπει καταρχάς να κατασκευάσουν αγωγούς πολύ περισσότερους και πολύ μεγαλύτερους από ό,τι είναι η πραγματική τους ανάγκη, γιατί εν καιρό θα ε, χρησιμοποιούν τους αγωγούς αυτούς και άλλες εταιρείες. Ε, και άρα χρειάζεται ένα είδος ε, κανονιστικής ρύθμισης, ένα είδος συντονισμού όλης αυτής της προσπάθειας και ε, συμμετοχή στο κόστος και το επιχειρηματικό μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Η έκθεση μου λοιπόν είχε σαν σκοπό να προωθήσει το CCS στην Ευρώπη και να φέρει κάποιες νέες ιδέες στο σύστημα. Ε, είδαμε πολύ ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες. Έχουμε τους πράσινους, την ΚΟΕ και τον Γκρότε, τα τρία G ε, δηλαδή που έκαναν όχι και τόσο επικοδομητικές ε, ε, τροπολογίες. Οι πράσινοι τουλάχιστον έχουν μια φιλοσοφία, επικοδομητική φιλοσοφία. Ενώ, πρόεδρε, για σας δεν ξέρω, δεν διαφωνούμε συχνά, ιδίως για θέματα κλιματικής αλλαγής, αλλά για αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα είμαστε κάπως αντίθετοι. Σε τελευταία ανάλυση δεν, σου αρέσει το CCS, α το πούμε ανοιχτά. Έτσι δεν είναι. Γιατί κοιτάζω τις τροπολογίες, όχι μόνο τις δικές, αλλά και άλλες τροπολογίες, που φαίνεται να λένε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα έπρεπε να έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στο να αποφασίσουν αν θα προωθηθεί όχι το CCS, και να δώσουν βοήθεια. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν τους, ε, συγγνώμη, συνάδελφοι που δεν τους αρέσει κανένα είδος ε, χρηματοδότησης, είτε άμεσης είτε μέσω πιστοποιητικών και σίγουρα δεν τους αρέσει η ιδέα ότι η Δοσία δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για βιομηχανικούς σκοπούς, αλλά ε, θα χρησιμοποιηθεί και για τις εκπομπές ε, καυσαριών από ηλεκτρο παραγωγούς σταθμούς. Δεν τους αρέσει το θέμα των αγωγών, δεν τους αρέσει η Κομισιόν να βοηθήσει να εντοπιστούν ε, πιθανή χώρη αποθήκευση στη Βόρεια Θάλασσα. Δεν τους αρέσει καν η αποθήκευση στη Βόρεια Θάλασσα, για προφανείς λόγους, μακριά από το σπίτι του καθένας και δεν θέλουν να δεχτούν ότι οι μακροχρόνιες προϋποθέσεις ε, βιωσιμότητας ε, που προβάλλουν οι ιδιώτες επενδυτές είναι υπερβολικές. Και σε τελευταία ανάλυση το κράτος μόνο θα πρέπει να αποφασίσει αν ένας τόπος είναι κατάλληλος για αποθήκευση. Και αν τελικά ε, υπάρχουν ε, προϋποθέσεις για δεκαετίες βιωσιμότητας, αυτό θα αποτρέψει κάθε ε, ιδιωτική επένδυση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και τόσο αρνητικές όλες οι τροπολογίες όπως φαίνονται εκ πρώτης όψεως και υπάρχει περιθώριο για επικοδομητικές διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς. Θα ξεκινήσουμε με τους πράσινους ε, για, τα ορυκτά καύσιμα και τους σταθμούς ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν θέλω να ε, έρθω σε αντίθεση μαζί σας. Μπορούμε να βρούμε τουλάχιστον μαζί με τους πράσινους, μια κοινή θέση που να λέει ότι υπάρχει ένας ρόλος για το CCS αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, βιομηχανικές εκπομπές και ούτε θα ε, τσακωθώ με τους ε, πράσινους για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Μπορούμε να βρούμε τη σωστή διατύπωση. Δεν νομίζω όμως, παρόλα αυτά, ότι μπορούμε απλώς να αγνοήσουμε το πρόβλημα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο λόγος που υπάρχει το CCS στην ατζέντα παγκοσμίω είναι διότι οι εκπομπέ διοξείδου του άνθρακα από άνθρακα και φυσικό αέριο αυξάνονται και δραματικά μάλιστα. Στην Κίνα, οι ε, ΙΠΑ ε, περνάνε από καύση άνθρακα σε καύση φυσικού αερίου, αλλά παραμένουν ε, στην καύση ε, ορυκτών καυσίμων. Όλα αυτά τα θέματα παρουσιάζουν μακροπρόθεσμα προβλήματα όσον αφορά την, ε, τον εφοδιασμό ε, σε ηλεκτρική ενέργεια. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πρόβλημα αυτό, ιδίως σε μια ε, περίοδο που οι εκπομπές αυξάνονται και πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την καύση άνθρακα και φυσικού αερίου. Δεν θα στεκωθώ όμω μαζί σας, όπως σας είπα, γιατί θέλω όσο γίνεται περισσότερο διακομματική υποστήριξη για να προωθήσουμε αυτή την ιδέα. Για να επανέλθω στη βιομηχανία, πριν κλείσω. βιομηχανία τσιμέντου το περασμένο μήνα ε, παρουσίασε ένα οδικό χάρτη για χαμηλέ εκπομπέ διοξείδου του άνθρακα. Λέει, άμα εφαρμόσουμε οποιαδήποτε τεχνική μπορούμε να ε, σκεφτούμε, μέχρι το 2050 θα μειώσουμε τις εκπομπές κατά 30%. Αν θέλουμε 80% αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς χωρίς το CCS. Η Ντάγμαρ μπορεί να λέει όχι, όχι, όχι, αλλά αυτό το λέει η τσιμεντοβιομηχανία. Δεν ξέρω αν η Ντάγμαρ μπορεί να εξηγήσει την τεχνολογία που υπάρχει και που η τσιμεντοβιομηχανία δεν μπόρεσε να σκεφτεί. Περιμένω να την ακούσω αυτή την εξήγηση. Λένε, με αυτά που ξέρουμε μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 30%, με το CCS κατά 80%. Αυτή είναι η διαφορά. Και το αναγνωρίζουν οι άλλες ομάδες μέσα στην Επιτροπή η βιομηχανία χρειάζεται το CCS αν πρόκειται να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σας λέω και πάλι το πρόβλημα της χημικής βιομηχανία στη Γερμανία. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. Ξεχάσετε τους αγωγού. Δεν είναι μόνο οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει να διαχωριστεί. Πρέπει να δεσμευτεί. Και αν δεσμευτεί, τι θα το κάνετε. Θα το βάλετε σε ένα ποταμόπλιο και θα το χύσετε στην ε, Βόρεια Θάλασσα. Για αυτό τώρα που ανησυχούν για την αντίδραση της κοινή γνώμης, το καταλαβαίνω, αλλά τα πράγματα είναι εύκολα για μένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει αντίρρηση. Όλοι, όλα υποστηρίζουν το CCS. Ρωτήστε κάποιον αν θέλει να είναι το σπίτι του πάνω από ένα πέτρωμα που δύο χιλιόμετρα από κάτω έχει θαυτεί το διοξείδιο του άνθρακα. Η Βόρεια Θάλασσα, σύμφωνα με τα τελευταία γεωλογικά ευρήματα, έχει αρκετά αποθέματα για όλα, όλες τις ποσότητες διοξείδου του άνθρακα από κάθε πηγή για 100 χρόνια για να αποθηκευτεί εκεί το διοξείδιο του άνθρακα για τα 100 επόμενα χρόνια και πρακτικά θα καλύψουμε όλες τις απαιτήσει για τους επόμενους αιώνες. Άρα μπορούμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες του, της κοινή γνώμης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά τελικά το θέμα είναι των κρατών μελών. Αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν το CCS, δεν θα συμβεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιβάλλουμε το CCS σε κανένα. Απλώ δεν θα εφαρμοστεί. Καμία εταιρεία δεν σκεφτεί καν να επενδύσει σε μια χώρα αν η κυβέρνησή τη, δεν υποστηρίζει θερμά ε, το πρόγραμμα αυτό. Άρα είναι τελικά και αποκλειστικά στο χέρι των κρατών μελών. Αν θέλουν το CCS να διαπραγματευτούν τις ρυθμίσεις πάνω στις οποίες θα βασιστεί και να ε, δώσουν και την απαραίτητη οικονομική βοήθεια. Απλώς ζητώ από τους συναδέλφους εδώ όταν υποβάλλουν τροπολογίες και σκέφτονται πώς θα ψηφίζουν, μην εμποδίζετε εκείνα τα κράτη-μέλη που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και να υιοθετήσουν αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Chris Davis, που έδωσες και ωραία παραδείγματα. Λοιπόν, η Σκιώδης τώρα. Η κυρία Γκροστέτ θα μιλήσει για την κυρία Γκαντίνη. Όχι, όχι, δεν ζήτησα τον λόγο. Κι όμως, κι όμως. Ναι, για την κυρία Γκαντίνη. Και ο κύριος Άντρες Κυρέλο Ροντρίγκες. Πρόεδρε, υπάρχει κάποιο σφάλμα. Εκ μέρους του εαυτού μου θα μιλήσω. Δεν έχω ευθύνη να μιλήσω για το σκιώδη συγητή από το ΕΛΚ. Εντάξει. Ε, αφού δεν έχετε ευθύνη για το ΕΛΚ, θα, η κυρία Ροντρίγκε για το, τους σοσιαλιστές, γιατί πρώτα θα μιλήσουν οι σκιώδει και μετά όλοι οι άλλοι. Ο κύριο Ροντρίγκε από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ. Σε όλε τι εκθέσει που εξετάζουμε εδώ έχουμε μεγάλε συζητήσει, διαφωνίε. Αυτή τη φορά το θέμα που εξετάζουμε δεν αποτελεί εξαίρεση. Και εδώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ πολιτικών ομάδων, μεταξύ χωρών, αλλά και μέσα στην ίδια πολιτική ομάδα. Αυτό αποτελεί και τον πλούτο εξάλλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω ποιο είναι ο στόχο τη έκθεση αυτή. Είναι να αναπτυχθεί η τεχνολογία δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε μεγάλη κλίμακα στι χώρε εκείνε που το επιθυμούν. Το είπε και ο κύριο αν το επιθυμούν οι χώρες θα το κάνουν, όχι αλλιώς. Υπάρχει βέβαια και το θέμα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, αλλά αυτά τα δύο, το CSS δηλαδή και ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, δεν είναι σε αντίθεση μεταξύ τους. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους αυτά τα δύο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα διασφαλίσουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωση συγχρόνως για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Συνεπώ. γι' αυτό εμεί υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες και ελπίζω να συμφωνήσουν όσο γίνεται περισσότεροι ευρωβουλευτές. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία γιατί η μεταλλουργία, η γεμική βιομηχανία κτλ φαίνεται να συμφωνούν. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας. Μπορεί να μην είναι τέλεια η λύση αυτή, αλλά είναι ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, κάποιες χώρες τουλάχιστον αυτές που θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όσο και αν μειώνονται τα ορυκτά καύσιμα, παρόλα αυτά θα αποτελούν πάντα το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού μείγματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ακούσαμε αυτό και το Μάρτιο του 2013 από την Επιτροπή που είπε ότι θα είναι απαραίτητο το σύστημα CSS για να ε, διατηρήσουμε την αύξηση της δημοκρατίας κάτω από τους δύο βαθμούς. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλες τις βιομηχανίες. Μέχρι τώρα πάντως διάφοροι μηχανισμοί έχουν αποτύχει δυστυχώς. Εξαρτώνται από την τιμή του άνθρακα και επειδή μειώθηκε η τιμή του άνθρακα σήμερα δεν υπάρχει κίνητρο για να γίνουν επενδύσεις στο σύστημα CSS. Άρα πρέπει να βρεθούν νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, η δημιουργία για παράδειγμα ενός ταμείου για τη βιομηχανική καινοτομία ή το θέμα των πιστοποιητικών είναι υποχρεωτικό για τους ε, εισαγωγείς, αλλά ενθουσιασμός προς το παρόν δεν έχει υπάρξει. Επιμένω ότι είναι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία θα, επιτρέ... θα αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν τον μηχανισμό δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στις χώρες τους ή όχι. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες οι οποίες θα αναλάβουν και το αρχικό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει πιο ενεργό ρόλο κυρίως για να προωθήσει την ανάπτυξη του συστήματος αυτού. Αλλά τα κράτη-μέλη παραμένουν με την δικιά τους ευθύνη. Αυτό που θέλω εδώ να υπογραμμίσω και με το οποίο δεν συμφωνούμε και πολύ με τον εισηγητή αλλά με άλλους ναι, είναι η ευελιξία στην ευθύνη που έχει κάποιος για την αποθήκευση. Γιατί δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό να έχουν την ευθύνη, ή να την αναλαμβάνουν ε, οι χώρες μέλη. Υπάρχει ένα πλαίσιο πάντως όσον αφορά την αποθήκευση για την ασφάλεια του συστήματος ε, αυτού. Είναι πάντως μια σημαντική πρωτοβουλία και η Επιτροπή μας θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα για τον ρόλο που μπορεί να παίξει το CSS. Ελπίζουμε να υπάρξει στήριξη είχαμε μέχρι τώρα, αλλά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στήριξη αυτή. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει μία πρόταση με την οποία να προωθήσει ακόμα περισσότερο το σύστημα CSS. Άρα είναι ουσιαστικό να μειωθεί το κόστος του και να αποτελέσει μια τεχνολογία η οποία εμπορικά να είναι βιώσιμη. Γιατί τελικά περί αυτού πρόκειται. Όταν ξεκινήσαμε με την, με την πρωτοβουλία αυτή, αυτό θέλαμε. Με τις τροπολογίες μας προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά τις διάφορες θέσεις και ελπίζω η έκθεση αυτή να αποβεί χρήσιμη και να μπορέσουν όλοι να ικανοποιηθούν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Κρίς ε, για την έκθεσή του, για τις αρχικές του παρατηρήσεις, ο κύριος Eichhout. Αρχίζω με κάτι αρνητικό προς εσένα, Κρίς, αλλά μετά θα δεις, θα πάρω πιο φιλικό τόνο. Ε, στην αρχή ρωτιόμουν, μα τι γίνεται με σένα, τέλος πάντων. Γιατί βλέπεις, ήσουνα πάντα κάποιος που στήριζε ε, το περιβάλλον το κλίμα. Και τώρα τελευταία βλέπουμε ότι έχει αλλάξει, έχει στραφεί προς την επίσημη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για το 30-30 και είσαι στη γραμμή του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει «Ε, η αγορά να αποφασίσει πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι δηλαδή η άποψη ότι η αγορά δίνει τον τόνο. Συγχρόνως όμως το Ηνωμένο Βασίλειο τι διαπιστώνει. Διαπιστώνει ότι δεν μπορεί η αγορά να τα προσφέρει όλα. Γιατί τη στιγμή που λέει ότι θέλουμε ένα στόχο, το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα αποφασίσουν οι αγορές, συγχρόνως λέει ότι για την πυρηνική ενέργεια θα δώσουμε 40 χρόνια. Άρα και αυτό το υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι και ο Κρίς. Επιπλέον λοιπόν τώρα για το CSS προτείνεις επιπλέον συγκεκριμένο στόχο για το 2020 στην έκθεση πρωτοβουλία σου. Συνεπώς εδώ δεν είναι οι αγορές. Οι αγορές δεν κάνουν αρκετά. Η... Το αποτέλεσμα της σου αυτής μπορεί να είναι ότι είσαι φιλόδοξος μεν, αλλά αυτό θες να το πετύχεις με τα πυρηνικά και το CSS. Ε, πώς γίνεται αυτό. Δεν θέλεις ε, ε, μείωση κατανάλωση ενέργειας, θέλεις το CSS και θέλεις και τα πυρηνικά. Ε, είναι περίεργο. Οπότε εδώ ανησυχώ για το δρόμο που παίρνουμε. Αλλά όπως σου είπα θα γίνω πιο φιλικός μετά, οπότε ξέφρασα την ανησυχία μου και τώρα περνάω στο πιο φιλικό σκέλος της παρέμβασής μου. Εδώ έχεις δίκιο. Κρίς, στο γενικότερο. Και εγώ πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα, αν δούμε τους μακροπρόθεσμους στόχους, δηλαδή έναν κόσμο που δεν θα χρειάζεται καθόλου CSS, εδώ ναι. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, η χαλιβουργία για παράδειγμα. Πολύ οξυγόνο χρειάζεται στην επεξεργασία και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δεσμεύσουμε το οξυγόνο είναι με το άνθρακα. Άρα καταλήγουμε στο διοξείδιο του άνθρακα. Εδώ δεν έχει να κάνει με την κατανάλωση ενέργειας, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να βγάλεις το οξυγόνο από το κοίτασμά σου. Συνεπώς, κάθε φορά που θα φτιάχνουμε, ε, ε, θα φτιάχνουμε χάλιβα, θα έχουμε σαν παράγωγο το διοξείδιο του άνθρακα, υποχρεωτικά. Εδώ χρειάζεται λοιπόν. Συνεπώ βλέπω την προστιθέμενη αξία του CSS σε τέτοιου είδου όμω εφαρμογέ. Αλλά το σύνολο του, της τεχνολογίας, ε, της ζήτησης για την τεχνολογία αυτή, μου θέτει το εξής ερώτημα. Γιατί εγώ να υποστηρίξω μια εφαρμογή την οποία τελικά θα χρησιμοποιήσει και θα επωφεληθεί από αυτήν η βιομηχανία διοξιδίου του άνθρακα. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει θέση για τέτοιου είδου βιομηχανίε στο μέλλον. Πρέπει να απαλλαγούμε για αυτέ. Οποιαδήποτε τεχνολογία λοιπόν παρατείνει την ζωή μια τέτοια τεχνολογία, για μένα πρέπει να καταργηθεί. Για τις χώρες μέλη το CSS είναι για να βοηθήσει αυτές τις βιομηχανίες διοξιδίου του άνθρακα. Συνεπώς, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το CSS είναι τόσο προβληματικό για μένα, γιατί κάποιοι εκφράζουν ανησυχίες, αλλά και εμείς ως πράσινοι, γιατί να υποστηρίξουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, ο οποίος τελικά θα έχει σαν αποτέλεσμα να επιζήσουν ακόμα περισσότερο οι βιομηχανίες που και είναι διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τελικά κρίς σε παρασύρουν λάθος φίλοι. Και μπορεί να συμφωνήσω μαζί σου στον αγώνα, όμως μόνο εάν τον κάνεις για μία εφαρμογή που δεν είναι οι βιομηχανίες που καίνε διοξίδιο του άνθρακα, αλλά άλλες εφαρμογές όπου ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ. Ενώ για την παραγωγή ενέργειας ξέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικέ. Ενώ για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές δεν υπάρχουν. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν λοιπόν πούμε ότι ναι, θα προωθήσουμε την τεχνολογία αυτή για να καλύψουμε και να καθησυχαστούν οι ανησυχίες μας όσον αφορά τις βιομηχανίες αυτές που αναπόφευκτα ε, ελευθερώνουν διοξίδιο του άνθρακα, ναι, αλλά αν είναι για, τις, ε, για τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, τότε όχι. Χρειαζόμαστε την τεχνολογία αυτή μόνο για κάποιες εφαρμογές. Αν με αυτό συμφωνήσουμε, καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα μπρος και ελπίζω να το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Κρις Ντέιβιντ για τη δουλειά που έκανε. Πολύ ενδιαφέρον που μου είπατε ότι η έρευνα έχει απαντήσεις γιατί πρόκειται για το μέλλον τα επόμενα 100 χρόνια. Ήδη γνωρίζουμε εμείς από το 2009 που άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις. Τότε διαπιστώσαμε το, το CCS είναι δυνατότητα. Τώρα επανερχόμεθα με πιο πολλές λεπτομέρειες και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα προγράμματα CCS, αυτά που αναφέρονται στην έκθεση, θα φροντίσουν να λειτουργεί σωστά η τεχνολογία και να είναι και βιώσιμα να είναι και εφαρμόσιμα γιατί είναι δαπανηρή αυτή η τεχνολογία. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία η οποία θα διατηρείται μόνο με επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Αυτές τις προτάσεις του Chris Davis και των άλλων θα τις υποστηρίξουμε ε, με βάση την ελευθερία επιλογής. Γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν και βέβαια την κοινή γνώμη. Δεν πρέπει να πιεσθούμε, να εξαναγκαστούμε, να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία CCS ή CSS. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες περιορισμού των ε, αερίων θερμοκηπίου χωρίς CCS. Κάποιες χώρες έχουν καταφέρει μερικά πράγματα Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ε, προκειμένου περί τεχνολογιών CCS και υπάρχουν οι σχετικές τροπολογίες που υπογραμμίζουν ότι το CCS μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ε, το πρόσχημα για να χρησιμοποιούνται άκρητα τα ορυκτά καύσιμα γιατί πάντα πρέπει να φροντίζουμε για εναλλακτικές εναλλακτικές στα ορυκτά καύσιμα και το λιγνίτι για να μην ε, ταλαιπωρούμε θα συνέχεια με το θέμα της χρηματοδότησης. Ευχαριστούμε. Η Φρανσουάς Γκροστέτ. Όχι, η Ντάγμαρ. Η Ντάγμαρ. Εγώ δεν θα ψακωθώ με την βιομηχανία και τα επιχειρήματά τους που τα ακούω 20 χρόνια. Η τσιμεντοβιομηχανία πάντως είναι γνωστή γιατί πάντοτε ε, τασόταν κατά των νέων τεχνολογιών. Πάντως νομίζω ότι η παρουσίαση έγινε με τρόπο εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Η Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Θέλω να στηρίξω τον Κρι Ντέιβι εγώ, γιατί το 2008 ήμουν εισηγήτρια, μάλλον συντάκτρια γνωμοδότησης για την Επιτροπή Βιομηχανία όσον αφορά τη δέσμευση και την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Είναι αλήθεια ότι τότε ήταν κάτι καινούριο για όλους μας και είχαμε αναποθέσει πολλέ ελπίδε στην τεχνολογία αυτή και στην χρηματοδότηση πιλωτικών προγραμμάτων κλπ. Σήμερα όμω έχουμε την διαπίστωση ότι έχουμε μείνει πίσω, η Ευρώπη έχει μείνει πίσω και είναι κρίμα γιατί αν η Ευρώπη πραγματικά ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα θα είχε μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για να εξάγει και την ε, γνώση της προς τα έξω γιατί υπάρχουν και άλλες η όπου χρησιμοποιείται ο άνθρακας Εβραίο και άρα η δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα είναι ένα σημαντικό θέμα και για αυτούς. Καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει το σύστημα αυτό να το χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε συστηματικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεδομένου ότι η επικουρικότητα είναι αρχή που πρέπει να τηρούμε και κάθε χώρα μέλος είναι ελεύθερη να αποφασίζει για την ενέργεια ε, που θα παράγει, η δέσμευση και η αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Γι' αυτό και η έκθεση του συναδέλφου μας Chris Davis μας επιτρέπει να ρίξουμε νέο φως στην υπόθεση αυτή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το ξανασυζητήσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθηση στο ζήτημα. Ξέροντας βέβαια ότι οι χώρες μέλη έχουν μεγάλη ευθύνη και κυρίως οι βιομηχανίες που κυρίως εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Άρα εδώ πρέπει να συνδυάσουμε τη χρηματοδότηση, να βρούμε το καλύτερο μείγμα, διότι η αγορά άνθρακα όντως δεν λειτουργεί σωστά σήμερα. Αλλά δεν είναι γι' αυτό που πρέπει να αποσιωπήσουμε το θέμα και να μην το συζητάμε. Κάθε άλλο. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή πραγματικά στηρίζω την έκθεση του Chris Davis Εννοείται θα εξετάσω όλες τις τροπολογίε προσεκτικά, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ρίξουμε νέο φως σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε. Όταν την πρωτοδιάβασα την έκθεση, θεώρησα ότι είναι καθαρή πρόκληση. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ε, η πρόθεσή σου, πάντως σπάνια μου συμβαίνει αυτό πολύ συχνά συμφωνούμε με τον Κρίς, όπως το είπε και εκείνος άλλωστε. Αλλά τώρα αυτή η τεχνολογία θεωρώ ότι είναι νεκρή η CCS. Και αν, ωραία ακούγονται στο χαρτί, θεωρητικά χρειάζεται το CCS στα χαλιβουργικία, στη, ε, στην τζιβεντοβιομηχανία και σε μονάδες παραγωγής που δεν έχουμε άλλη δυνατότητα ε, για να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά έτσι όπως είναι φτιαγμένη η έκθεση, έτσι όπως ε, ε με τα ορυκτά καύσιμα, εκεί υπάρχουν εναλλακτικέ και πρέπει κάποιος να μου το εξηγήσει να το καταλάβω. Γιατί το βαθμό αποτελεσματικότητας μιας μονάδας παραγωγής ε, ενέργειας πρέπει να μειωθεί για να γίνεται η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, για ένα νέο εργοστάσιο. Νομίζω ότι το CCS εδώ ε, είναι η τελευταία εναλλακτική. Μόνο αν δεν υπάρχει άλλη θα χρησιμοποιείται. Ε, εκεί που υπάρχουν εναλλακτικέ στην παραγωγή ενέργειας πρέπει να αξιοποιούνται. Να είμαστε προσανατολισμένοι στο καινούριο. Μιλήσαμε και για το εμπόριο των, ε, και τα δικαιώματα των αερίων. Τι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από όλα αυτά. Θυμήθηκα τη δεκαετία του 90 που δεν ξέραμε ακριβώ πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Η τιμή ε, άνθρακα μπορεί να μας βοηθήσει για να χρηματοδοτήσουμε άλλα πράγματα. Ε, εξοπλισμοί, σύγχρονοι μέθοδοι ε, ηλεκτροδότησης των δρόμων. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλά που θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας. Βέβαια, αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα των κρατών μελών. Αν δούμε όμως τις επενδύσεις τα επόμενα 20 με 40 χρόνια, θα πρέπει να σκεφτόμαστε από το τέλος προς την αρχή. Το ευρώ που θα δώσω θα είναι δεσμευμένο για τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια. Πού πρέπει να μας οδηγήσει το ταξίδι μας και τι πρέπει να γίνει ούτω ώστε να πετύχουμε ε, ένα στόχο 70-80%. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει ε, επένδυση σωστή από άποψη κόστους ωφέλους, αλλιώς η αποδοχή ε, θα είναι προβληματική Στη χώρα μου αναφέρθηκε ε, ένα πείραμα που έγινε με την ενεργειακή στροφή και όταν οι τιμές ενέργειας ε, φτάσουν πολύ ψηλά, τότε η αποδοχή θα γίνει μηδενική και θα υπάρξει ε, αντιστροφή από αυτή την ενεργειακή καμπή και την σχετική πολιτική. Δεν είναι όλα λάθος όσα λέει η έκθεση, όχι, το ομολογώ, το παραδέχομαι, κάποια ε, με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά με την πρώτη ματιά ένιωσα ότι η έκθεση αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ε, και αυτό δεν οφείλεται στην πολιτική των τριών G που είπες, αλλά τη βαθιά μου πεποίθηση ότι πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές ε, όταν πρόκειται να βγάλουμε στην αγορά αυτή την τεχνολογία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να ε, βγάλουμε κάτι που δεν θα το μιμηθεί κανείς, δεν θα το θέλει κανείς, θα πρέπει να έχουμε ένα βαθμό οριμότητα στην αγορά για να το βγάλουμε και νομίζω ότι και εγώ μηχανικός είμαι και στην εκλογική μου περιφέρεια αυτές τις αντιδράσεις μπόρεσα να παρακολουθήσω και να κρίνω. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή μαζικά, δεν έχουμε φτάσει σε σημείο τέτοιο ώστε μαζικά να εφαρμόσουμε μια τέτοια πολιτική. Ε, την κυρία Κλάς μου φαίνεται ότι την προκάλεσα να λάβει το λόγο. Όχι, όχι δεν με προκαλέσατε κύριε Πρόεδρε, με προβληματίσατε. Γιατί είναι αξιοσημείωτο αυτό. Είχαμε τα πιλωτικά προγράμματα και τις εκθέσεις που, για τα πρώτα στάδια, αλλά δεν προχωρούν και υπάρχει μεγάλος φόβος γιατί δεν βρίσκουμε και μια μονάδα παραγωγής. Από την άλλη, και έχω παρακολουθήσει τη συζήτηση, βλέπω ότι δεν μπορεί να ε, ε, αυξήσουμε την χρήση του άνθρακα γιατί θα το θάβουμε στη γη. Από την άλλη, Μιλήσατε και για τη χαλιβουργία και για την τζιμετοβιομηχανία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ώστε να αρχίσει να χρησιμοποιείται η τεχνολογία, όχι όμως σε ευρεία κλίμακα, σε κάνα δυο μονάδες παραγωγής και να υπάρχει η δυνατότητα της δοκιμής να το δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Έτσι ενδεχομένως θα διασκεδαστούν και κάποιοι φόβοι που υπάρχουν. Μου φαίνεται ότι έτσι το εννοεί και ο Chris Davis. Να το δούμε να γίνει ένα πιλωτικό, να το υπομιστούμε όλοι, να το παρακολουθήσουμε καλά και να μην είναι ευρεία η εφαρμογή. Να είναι δηλαδή ένα που να το δούμε καλά. Έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση αυτό, το είπα και στην αρχή, θα δώσω και στον Chris Davis τον λόγο να απαντήσει και η Κομισιόν επίσης. Τώρα, τα έσοδα από το εμπόριο των εκπομπών χρησιμοποιούνται από τον κλάδο για την προώθηση και άλλων τεχνολογιών. Αν αφαιρέσουμε κάποια κονδύλια από εκεί θα πρέπει να τους το πούμε. Ε, ας πούμε οι δήμοι κοινότητε στη χώρα μου περιμένουν από το πρόγραμμα αυτό κάποια χρήματα γιατί υπάρχει υποχρηματοδότηση εκεί. Περιμένουν λοιπόν να πάρουν λεφτά για να φωτίσουν τους δρόμους με λιχνίες LED. Ε, να έχουν έτσι ένα χρηματοδοτικό περιθώριο οι δήμοι και οι κοινότητες. Δεν μπορεί να πάρουμε απόφαση να βάλουμε όλα τα λεφτά στην τεχνολογία CCS με αβέβαιη έκβαση. Δεν συνεχίζω όμως, θα δώσω στην Κομισιόν το λόγο και μετά στον Chris Davis για να κλείσει και να ε, αντιδράσει με λάκτισμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σήμερα εδώ και επιθυμεί να λάβει το λόγο να μιλήσει. Α, δύο είναι μάλιστα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η Κομισιόν καλωσορίζει θερμά την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σχετικά με την σημασία και το μέλλον του CCS στην Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή είναι πραγματικά πολύ επικαιρή και σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δουλειά που έχει αναλάβει η Κομισιόν. Μετά από δύο δημόσιες ε, διαβουλεύσεις που ξεκίνησε φέτος το Μάρτιο, η Κομισιόν για το 23ο πλαίσιο για το κλίμα και ε, τις σχετικές συζητήσεις ε, συνεχίζονται οι σχετικές διαβουλεύσεις στο εσωτερικό της Κομισιόν. Όπως ξέρετε, η Λευκή Βίβλος που θα δημοσιευτεί του χρόνου θα θέσει κάποιους προσανατολισμούς όσον αφορά την πολιτική μας και το CCS πιστεύω ότι θα έχει τη θέση του εκεί μέσα. Και η θέση αυτή θα σχετίζεται με τους συνολικού στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και με τους στόχους για το 2030 και 2050 ε, των κρατών μελών. Βεβαίως, ε, όπως υπόθηκε, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για να ε, επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα και κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποφασίσουν το κατά πόσο θα έχουν CCS στα εδάφη τους. Και βλέπουμε πολύ διαφορετική εικόνα στα διάφορα σημεία της Ευρώπης. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι το CCS μπορεί όντως να παίξει έναν, ε, έναν ε, σημαντικό ρόλο στην ε, απομάκρυση από τον άνθρακα της Ευρώπης στο μέλλον μαζί με μέτρα αποδοτικής χρήσης ενέργειας και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης δεν θα ξεχνάμε ότι η τεχνολογία CCS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος πηγών διοξιδίου του άνθρακα. Όχι μόνο για τον άνθρακα δηλαδή, αλλά υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και για άλλους βιομηχανικούς κλάδους, όχι μόνο για την ηλεκτροπαραγωγή. Και σε κάποια είδη βαριάς βιομηχανίας όπως ε, και χαλιβουργίες. Το CCS θεωρείται ότι είναι η μόνη τεχνολογία που μπορεί να δεσμεύσει τουλάχιστον το 90% των εκπομπών από τους μεγαλύτερους, ε, μεγαλύτερες πηγές εκπομπών στον κόσμο. Το CCS δεν είναι αναγκαστικά σε ανταγωνισμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορεί να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ε, μπορεί να υποστηρίξει το CCS της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξασφαλίζοντας ε, την συνέχεια της του ενεργειακού ε, φοδιασμού να ε, οδηγήσει σε μεγάλες μειώσεις ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πολύ μεγαλύτερες από ότι οι ανανεώσιμες πηγές από μόνες τους. Άρα ε, ένας συνδυασμός τεχνολογιών θα είναι απαραίτητος για να επιτύχουμε τους στόχους μας για απομάκρυση από το, τη χρήση του άνθρακα. Φυσικά Όλοι ξέρουμε ότι το οικονομικό μέρος του CCS πρέπει να βελτιωθεί. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν το διοξίδιο του άνθρακα θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εμπορίας σαν ένα οποιοδήποτε αγαθό. Και επίσης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να ενθαρρύνει ε, έργα επίδειξης του κόστους και της αποδοτικότητας της τεχνολογίας του CCS. Αν θα μου επιτρέπατε να προσθέσω κάτι στα σχόλια που έγιναν σήμερα, λέει, ο άλλος εκπρόσωπος της Κομισιόν, για την, ε, τα έργα επίδειξη στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη δύο ταμεία που οργάνωσε, ε, θέσπισε η Κομισιόν. Το ένα είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης και το άλλο είναι το πρόγραμμα ε, που συνεχίζεται ακόμα το NER 300. Πιστεύουμε ότι το NER 300 θα έχει σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα έργο επίδειξης και εφαρμοσιμότητας του συστήματος στην Ευρώπη και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για το CCS. Όπως είπε η συνάδελφος, το CCS θεωρείται ακόμα μία από τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, ε, την Ευρώπη να πιάσει τους στόχους του 2050. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ελπίζουμε ότι η Λευκή Βίβλος που θα δίνει τους προσανατολισμούς για το 2030 θα ξαναφέρνει στην επικαιρότητα το ε, πρόγραμμα αυτό. Κάτι τελευταίο σχετικά με τον ορίζοντα του 2020 και το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την υπάρχει εκεί μια ε, διάταξη, μια πρόβλεψη για την πρόθεση αυτής της τεχνολογίας, για μείωση του κόστους, για καλύτερη κατανόηση του πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο Θέλω για αυτά που άκουσα από τον Μπάσκετ την τάγμαρ να αντιδράσω έντονα, γιατί είναι κατηγορίες. Τι λέει, λέει μας ότι εγώ έχω εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις μου και ότι έχω αλλάξει την άποψή μου για τα περιοδικά και τα λοιπά. να κατά για χρόνια. Αλλά δεν εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Τι να κάνουμε, αυτό το αναγνωρίζω. Υπάρχουν βέβαια ενεργά απόβλητα, βεβαίως, γι' αυτό. Οπότε εσείς δεν ξέρω με προκαταλήψεις ε, συζητάτε. Είμαι έξαλλος. Όσο για την βιομηχανία άνθρακα. Μα οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Θέλουν να καταρρεύσει το σύστημα. δεν κάνουν τίποτα για να δείξουν την ε, χρησιμότητα που έχει το σύστημα. Τώρα, Ντάκμαρ, ναι, έχουμε εκλογέ την επόμενη χρονιά και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι φιλελεύθεροι που είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε τον κύριο Μάτ εδώ από το Independence Party που θα πει ότι όλοι οι ξένοι Ευρωπαίοι θα έρθουν ε, σε εμά και θα μας καταστρέψουν. Ωραία. Να πάω κι εγώ λοιπόν στην προεκλογική εξαρτήτα στην Τάκμαρ και να πω χρειαζόμαστε το σύστημα αυτό δέσμευσης και αποθήκευσης. Για τα σχόλια των υπολείπων, Ροντρίκης, Γκροστέτ κλπ όσον αφορά το στόχο. Αν χρειαζόμαστε στόχο για το 2020 για το CSS. Μα κυρία Κρουστέτ, έχουμε στόχο. Τον έθεσε το Συμβούλιο το 2007. 12 έργα CSS που να λειτουργούν το 2050. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν έχουμε κανένα, δεν έχει αρχίσει κανένα από τα 12. Οπότε εντάξει, το στόχο το ξέρουμε και για τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό που θέλω εγώ είναι κάτι να γίνει ότι υπάρχουν προτεραιότητες και θα αρχίσουν να λειτουργούν κάποια από αυτά τα προγράμματα. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα, αλλά η προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι η ίδια που τα κατά το παλθόν. Πρέπει να είναι να μπει η βιομηχανία πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και θα αναπτύξουμε μια τεχνολογία πολύ σημαντική για όλους. Προς το παρόν, έχουμε μια πολιτική οι οποίοι, μάλλον δεν έχουμε καθόλου πολιτική για κίνητρα προ τη χημική, την τσιμετοβιομηχανία ή οποιαδήποτε άλλη ώστε να προτείνουν προγράμματα, έργα. Ούτε έχουμε κανέναν από τους διάφορου κλάδους που να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πει ναι, να συνεργαστούμε, να έχουμε από κοινού ένα πακέτο. Οπότε κάνω έκκληση στι βιομηχανίε αυτές να συμβρεθούν για κέρδος, να μην υπάρχει απώλεια. Χρειάζονται όμως επιδοτήσεις, χρειάζεται βοήθεια. Όμω πρέπει να έρθουν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να πούνε θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναπτύξουμε μια στρατηγική για να προωθηθεί η τεχνολογία αυτή και θέλουμε να την αναπτύξουμε πριν έχουμε μείνει τόσο πολύ πίσω όπως διάφοροι άλλοι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 27 και 28 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια θα πάει Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2014. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προχωράμε τώρα. Σημείο 6. Το θέμα της Μαγιότ. Εγώ είμαι ο συγγητής. Για το, τη Μαγιότ μιλήσαμε στο προηγούμενο Στρασβούργο στην ε, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι από πρώτη πρώτου άλλαξε το καθεστώς και χρειάζονται κάποιες ε, έκτακτες ε, εγκρίσεις για περιβαλλοντικά πρότυπα Πήραμε γνωμοδότηση της Επιτροπής, της Νομικής Επιτροπής. Δεν δεχόμαστε να μην υφίσταται πια η συναπόφαση, αλλά να έχουμε μόνο διαβούλευση. Ε, κάποιοι συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες με διπλή νομική βάση. Τώρα έγινε προπόντιο διαμέρισμα η Μαγιώτ πρέπει να δούμε μήπως αποδυναμώνεται η θέση του Κοινοβουλίου. Εμείς πρέπει να δράσουμε ευσυνείδητα και επειδή ε, υπάρχουν κάποιες χρονικές πιέσεις βάλαμε εμβόλυμα μια συνεδρίαση στις 14 Νοεμβρίου εκτάκτως 9 η ώρα το πρωί. Ελπίζω να έχουμε όλη πλήρη ενημέρωση της κατάστασης αλλά και της ε, νομικής βάσης. Εγώ θα βάλω τη νομική υπηρεσία να μας τα ξαναπεί. Οι Λεπάζ, Λεόγκ, Φράγκο, Μπρόγκα, Πανιό κατέθεσαν τροπολογίες σχετικά, δηλαδή με τη διπλή νομική βάση. Δηλαδή όλοι είναι Γάλλοι και διαπαραταξιακά συμφώνησαν σε μια γραπτή, γραμμή πλεύσης. Δυστυχώς όμως δεν εκπροσωπούνται εδώ από κανέναν. Πάντως θα συζητήσουμε το ε, θέμα και αργότερα. Τώρα, ε, για να αρχίσουμε τη συζήτηση, δεν βλέπω σκιώδης. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη, παρακαλώ. Εγώ έχω ένα μήνυμα από το σκιώδη της ομάδας ECR. Και το μήνυμα είναι απλό. Το θέμα είναι εθνικό, είναι γαλλικό και δεν θεωρεί να, ότι πρέπει να ανακατευτούμε εμείς. Κατόπιν τούτου θεωρεί ότι το νησί είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει επίσης να καλύπτεται και από την ενωσιακή νομοθεσία. Φινίτο. Ε, τελείωσα. Μάλιστα, ε, τελειώσα. Άλλος κανείς ζητεί το λόγο. Η Κομισιόν παρακαλώ. Α, η κυρία, Γκροσ... ε? κυρία Γκροστέτ. Είναι γεγονός ότι δεν είχα κάνει τροπολογίας με τους Γάλλους συναδέλφους. Η τότε έγινε ένα ε, διαμέρισμα γαλλικό, άρα εφαρμόζεται η κοινωτική νομοθεσία, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος για να οργανωθούν όλα αυτά. Ε, δεν είναι καθόλου πρόφανες όταν γνωρίζει κανείς την κατάσταση στη Μαγιότ ε, πώ θα καταφέρει από μια μέρα στην άλλη να ε, συμμορφωθεί με το κοινοτικό κεκτημένο. Εγώ δεν έχω κάνει διερευνητική επιτροπή ως εισηγητής, αλλά μου είπαν ότι έγινε το 101ο υπερπόντιο διαμέρισμα πλέον, η Μαγιότ. Η Κομισιόν παρακαλώ, ας μας διευκρινίσει ποιος ε, θα λάβει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. We would Θα θέλαμε να κάνουμε μια δήλωση πολύ σύντομη για την νομική βάση και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου για τα θέματα ε, ουσίας. Είναι περιττό να πούμε ότι είμαστε κατά της διπλής νομικής βάσης για ένα πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, πρόκειται για ένα ενιαίο αντικείμενο και αν όπως λέει η Επιτροπή Γιούρι είχε δίκιο η Κομισιόν που χρησιμοποίησε την κανονική νομική βάση, δηλαδή την τομεακή νομική βάση που ισχύει στους διάφορους επιμέρους τομείς, τότε για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο μια πρόσθετη νομική βάση δεν μπορεί να είναι κάτι το σωστό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. επιλέξαμε την κανονική νομική βάση, να σας το υπενθυμίσω αυτό, γιατί σε οποιαδήποτε περιοχή μπορεί να κάνει κανείς ε, γεωγραφικές διαφοροποίησεις όταν αυτό δικαιολογείται. Εδώ θεωρούμε ότι δικαιολογείται κάτι τέτοιο και κάνουμε προτάσεις με βάση την κανονική νομική βάση που περιλαμβάνει και στην απόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν αυτό είναι σωστό, τότε το άρθρο 349 είναι λάθος. Είναι λάθος σαν α, η μόνη νομική βάση, αλλά είναι εξίσου λάθος και σαν μια πρόσθετη νομική βάση. Το ίδιο πράγμα δεν μπορεί να έχει δύο ονόματα. Και δίνω τώρα το λόγο ε, στον συνάδελφο για τα θέματα ουσίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τοποθετηθώ για ορισμένα σημεία ε, της πρότασης ε, όπου υπάρχουν προτάσεις για αλλαγές σε σχέση με τον ε, αριθμό ισοδύναμου πληθυσμού και ε, επίσης η Κομισιόν ε, πρότεινε να λάβουμε υπόψη μας τις πληροφορίες που μας ήρθαν από τη Γαλλία και η Κομισιόν για το λόγο αυτό σκέφτηκε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αν λάβουμε υπόψη αυτές τις οδηγίες και άλλες οδηγίες αντιφατικές σε σχέση με το περιβάλλον. Αλλά χωρίς την εφαρμογή αυτών των οδηγιών, ε, οι οδηγίες για το νερό ή για, το, για τα ύδατα δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ουσιαστική η εφαρμογή αυτών των οδηγιών για την κοινωνική, την περιβαλλοντική, την ανθρώπινη ανάπτυξη, αν μπορώ να πω, του πληθυσμού. Η Κομισιόν λοιπόν μπορεί να κάνει κάποιες ε, δηλώσεις σε σχέση με τις τροπολογίες που προτείνει το Κοινοβούλιο που κατά τη γνώμη μας έρχονται αντίθετα με τη λογική της οδηγίας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες που δεν προέρχονται από την οδηγία και αυτό ισχύει για κάποιες τροπολογίες που χρησιμοποιούν τον όρο municipalities, δήμοι δηλαδή, αντί για οικισμοί, αυτό είναι αντίστοιχο με το πνεύμα της οδηγίας, ή κάποιες άλλες τροπολογίες που αναφέρονται στον αριθμό του ισοδύναμου πληθυσμού που πρότεινε η Κομισιόν. Αν ο γενικός στόχος του να έχουμε το 70% της ρήπανσης ε, που παράγεται στη Μαγιότ ε, το 70% ε, να υφίσταται επεξεργασία μέχρι το 2020, αν αυτός είναι ο στόχος, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα, κατά τη γνώμη της Κομισιόν πρέπει να μείνουμε συνεπείς με αυτούς τους στόχους και δεν θα πρέπει να θέτουμε υπό ε, την αρχή πρόταση της Κομισιόν που μιλάει για οικισμούς 10.000 ε, ισοδύναμου πληθυσμού. Και όλα αυτά ε, με σεβασμό προς ορισμένες προτάσεις που φαίνεται να θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο και που συμβάλλουν στο να διευκρινιστούν οι στόχοι που έχει θέσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ζητεί από ό,τι βλέπω άλλο το λόγο για να πει για τη νομική βάση. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ε, παλέψουμε για τη διατήρηση της συναπόφασης. 27-28 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε, ε, Νοεμβρίου συγγνώμη, και 14, 14 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. 14. Και προγραμματίζεται για να πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και να ψηφιστεί εκεί. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, και τώρα να καλέσουμε μέσα τον προσκεκλημένο μας. Καλωσορίζω θερμά τον Υπουργό Υγείας της Προεδρίας. Στην πρώτη παρουσίαση του αναφέρθηκε ότι έχει στενές επαφές με το Κοινοβούλιο και συχνά επιθυμεί ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα που εκκρεμούν. Πράγματι, ε, όλο αυτό το διάστημα ε, ε, έκανε αυτό που είχε πει. Μπορούμε λοιπόν να σας δώσουμε το λόγο για να μας ενημερώσετε και μετά θα λάβουν το λόγο και οι συνάδελφοι για ερωτήσεις. Ευχαριστώ Ματίας. Αξιότιμε πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να σας συναντήσω για μια ακόμη φορά και να σας παρουσιάσω μια ενδιάμεση έκθεση ε, στα θέματά μας ε, από τη Λιθουανική Προεδρία. Μόνο σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να συνεχίσουμε. Έτσι δημιουργείται θετικό δυναμικό πνεύμα ε, το οποίο ελπίζω να ε, κρατήσει το επόμενο δίμηνο και ε, πραγματικά η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τέλεια. Ε, έτσι λοιπόν θέλω να συζητήσουμε μαζί τι καταφέραμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα. Συνεχίζω στα αγγλικά. Δεν ήρθα εδώ μόνο για να απαντήσω σε ερωτήσεις, αλλά να πάρω τις δικές σας απόψεις, τις ε, ιδέες σας, ε, τις προοπτικές σας. Είναι πολύ σημαντικός ένας τέτοιος διάλογος αφού είναι και περίπλοκα τα θέματα που πρέπει να λύσουμε μαζί. Όπως ξέρετε τώρα ε, συζητάμε με πολύ δραστηριό τρόπο το θέμα των σύγχρονων διώσιμων ε, συστημάτων υγείας ε, προσάρμοστων και το πώς θα συζητηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στην ομάδα εργασίας. Θα πρέπει να δούμε την υγεία στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική χρήση των διορθωτικών ταμείων για επενδύσεις στην υγεία, ε, αποτελεσματική χρήση φαρμάκων, ε, μοντέλα ε, ε ολοκληρωμένης φροντίδας και καλύτερη νοσοκομιακή περίθαλψη και διαχείριση ε, παρακολούθηση τη αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στην υγεία. Όμως ε, τα συστήματα, τα σύγχρονα για την υγεία και μια σύγχρονη πολιτική δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να είναι μόνο ε, μια δαπάνη που δεν δημιουργεί αξία, αλλά θα είναι αναγνωρισμένος παράγον που συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση θα μειώνει την φτώχεια, θα αυξάνει την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Η μείωση των ανισοτήτων είναι κλειδί για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Υπενθυμίζουμε τη σημασία της υγείας σε όλες τις πολιτικές και τις αρχές αλληλεγγύης όπως και η συμμετοχή άλλων τομέων και η στενότερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα είναι παράγοντες κλειδί στην σύγχρονη πολιτική υγείας. Αυτές οι ιδέες έχουν συζητηθεί αλλά πρέπει να συζητηθούν κι άλλο σε πολλά ε, φόρα και θεωρώ ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου να σας παρουσιάσω τώρα τα αποτελέσματά μας σε σχέση με τις σημαντικότερες νομοθετικές προτάσεις. Καταρχήν για τον καπνό. Πρώτα να σας συγχαρώ για την καλή δουλειά που κάνατε για την οδηγία για τον καπνό και να συγχαρώ και την εισηγήτρια Λίντα Μακάβαν που άρχισε τον τριμερείς διαλόγους. Η Λιθουανική Προεδρία χαιρέτησε την ψήφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που απέδειξε ότι οι στόχοι των δύο συνομοθετών ταυτίζονται και τα σχέδια τροπολογιών του Κοινοβουλίου και η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση σε από, από πολλές απόψεις. Εμείς τώρα θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις πρώτες διαπραγματεύσεις, ε, ε, τις διαπραγματεύσεις πρώτης ανάγνωσης πριν από το τέλος του 2013, οπότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια οδηγία για τα προϊόντα καπνού που επίσημα θα εγκριθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Συμφωνώ με το επιχείρημα του Κοινοβουλίου ότι αυτή η οδηγία είναι σημαντική διότι εφαρμόζει τη σύμβαση πλαίσιο του ΠΟΗ για τον έλεγχο του καπνού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πίσω από τη Βραζιλία, τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία και κάποιες άλλες χώρες. Και είναι κοινό μας καθήκον να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Ε, ανακτώντας την παγκόσμια ηγετική θέση στο θέμα ελέγχου καπνού. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να διαπραγματευτούμε ακόμα, όπως ε, το θέμα των συστατικών, των ηλεκτρονικών τσιγάρων, διασυνοριακών πωλήσεων, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο βασικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι δεν θα αρχίσουν να καπνίσουν. Να καπνίζουν ενώ άλλοι θα σταματήσουν ή θα μειώσουν το κάπνισμα. Γι' αυτό ε, στηρίζομαι πολύ στην κατανόηση και την στήριξή σας ε, για να συμφωνήσουμε από κοινού σε αυτή την ε, νομική πράξη, νομοθετική πράξη. Δεν πρέπει να θυσιάσουμε τους βασικούς στόχους για υπερτεχνικών λεπτομεριών όπου μπορούμε να βρούμε συμβιβαστική λύση. Κλινικές ε, δοκιμές για τις φαρμακευτικές ουσίες. Αυτό είναι σημαντικό για να αναπτύξουμε νέα φαρμακευτικά προϊόντα και καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα φαρμακευτικά προϊόντα προς όφελος των Ευρωπαίων ασθενών και για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνοντας έρευνα και καινοτομίες. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ευρώπη αν θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες της Ένωσης πρόσβαση σε καλύτερα φαρμακευτικά προϊόντα και να διατηρήσουμε ε, μια στιβαρή φαρμακευτική βιομηχανία η οποία θα δημιουργεί υψηλής εξειδίκευσης θέση εργασίας. Ο κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές ε, πληρεί το στόχο αυτό, γιατί ενθαρρύνει την κλινική έρευνα στην ε, Ένωση, μειώνοντας το διοικητικό φόρτο, ενώ διατηρεί ε, προστασία σε υψηλό επίπεδο. Το... Η εντολή από την Κορεπέρ δόθηκε στην Προεδρία στις 30 Οκτωβρίου και οι διαπραγματεύσεις το, Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο θα αρχίσουν 6 Νοεμβρίου. Χρειάζεται μια ισορροπημένη προσέγγιση ορθολογική για να έχουμε κοινή συμφωνία πάνω στον κανονισμό. Τονίζω ότι δεν πρέπει να δαπανίσουμε πολύ χρόνο πάνω στα τεχνικά θέματα, αλλά να εστιάσουμε στην έγκαιρη έγκριση αυτής της νομοθετικής πράξης. Η Λιθουανική Προεδρία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχει συμφωνία επί της πρότασης, επειδή τα περισσότερα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει την ε, στεναρή τους ετοιμότητα να δουλέψουν για ε, γρήγορη έγκριση αυτή της νομοθετική πράξη, που είναι τόσο σημαντική. Υπογραμμίζω και πάλι ότι αυτός ο κανονισμός είναι τεράστια σημασία για ασθενείς, με ακαδημαϊκή έρευνα και τη βιομηχανία. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην εισηγήτρια Γκλένις Βίλμοντ και την ομάδα της για τη σκληρή δουλειά που έκαναν για να προετοιμάσουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλω να, τη, να διασφαλίσω ότι προσβλέπουμε σε μια μελλοντική συνεργασία ακόμα πιο στενή τώρα που θα επιδιώξουμε συμφωνία πάνω σε αυτή τη σημαντική νομοθετική πράξη. Τέλος να πω ότι η Λιθουανική Προεδρία εργάστηκε σκληρότατα για να ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να πούμε ότι μεγάλη πρόοδος επετέφθη ε, στην εξέταση του Συμβουλίου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα θέλω να καλέσω όλα τα μέρη να εργαστούν επικοδομητικά από κοινού και ελπίζομαι ότι αυτή η σημαντική νομοθετική πράξη θα συμφωνηθεί επί Λιθουανικής Προεδρίας. Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και προϊόντα. Η Προεδρία έχει αναλάβει δέσμευση να επιτύχει τη μέγιστη πρόοδο επί δύο προτάσεων για κανονισμούς στη ιατροτεχνολογικά και στη διαγνωστικά in vitro. Ε, η πρόταση επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς που υπάρχει τώρα για την αδειοδότηση των ιατροτεχνολογικών για τα κράτη-μέλη πρέπει να εξετάσουν πολύ προσεκτικά τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα αυτά στο υφιστάμενο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλά τεχνικά θέματα που έχουν ρυθμιστεί σε εθνικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια δύο οδηγιών θα πρέπει τώρα να συμφωνηθούν σε επίπεδο ένωσης. Αυτό σημαίνει μακράες συζητήσεις πιο μακρέ συζητήσει επί του νέου συστήματο εποπτείας και επιτήρηση των ιατροτεχνολογικών ε, βοηθημάτων που προβλέπονται από αυτού του κανονισμούς. Ο στόχο τη Λουθανική Προεδρίας είναι ε, να προχωρήσει γρήγορα. Όμως η πρόοδος δεν είναι ταχεία. Γι' αυτό θέλουμε να αρχίσουμε συζητήσεις με συναδέλφους για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Ε, ε, να υπάρξουν φρέσκες ιδέες για περαιτέρω πρόοδο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, εισηγήτρια Ντάγμα Ροτμπέρντε και τον εισηγητή για την πρόταση για τα in vitro, τον Dr. Πέτερ Λίζε, για τη στήριξη και την ενεργό θέση τους. Ε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί τους για να βρούμε πιθανές λύσεις για να υπάρξει πρόοδος και επί ελληνικής προεδρίας. Φάρμακο επαγρύπνηση ε, και ο κανόνας για τα τέλη τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πρακτική εφαρμογή νέας, εφαρμο... και τη χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων φάρμακο επαγρύπνησης θα γίνεται και από τους εθνικούς φορείς και από την ΕΜΕΑ. Εμείς ελπίζουμε ότι θα αρχίσουμε τριμερείς διαλόγους. Στηριζόμεθα, στις... υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας γιατί αυτή η νομοθετική πράξη πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν για την καλύτερη εφαρμογή των νόμων φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα δουλέψουμε στενά με την εισηγήτρια Λίντα Μακάβαν για να έχουμε συμφωνία σε αυτό το σημαντικό φάκελο και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσουν τη θέση τους στο ταχύτερο δυνατόν. Αλλά νομοθετήματα. Ε, το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία για την ανάπτυξη ε, είναι πολύ σημαντική για την νέα αυτή δημοσιονομική περίοδο. Πρέπει να εγκριθεί ε, Τώρα πάμε να λύσουμε κάποια ακόμα εκρεμή θέματα, συνεργαζόμενοι με Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθεί το πρόγραμμα. Συνεχίζονται οι συζητήσει για τη λεγόμενη διαφάνεια, ε, συμπερίληψη δηλαδή ε, των φαρμάκων στο σύστημα επιστροφής, ε, ε τιμολόγησης κλπ. Ε, πρέπει να ελπίζουμε να οργανώσουμε μία ακόμα συνάντηση της ομάδας εργασίας για αυτό το θέμα, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ετοιμότητα των άλλων κρατών μελών που θα πρέπει να συμφωνήσουν σε επισύμβιβαστικών μου προτάσεων και αυτό ακόμα δεν έχει οριμάσει. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, επιτρέψτε μου να σας ε, παρουσιάσω τα, ε, τις επόμενες εκδηλώσεις του προγράμματος της Προεδρίας και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε. Εκδηλώσεις της Προεδρίας αντικατοπτρίζοντας την, ε, απηχώντας την σημασία των προβλημάτων ψυχικής υγείας, η Προεδρία ε, διοργάνωσε υψηλού επίπεδου διάσκεψη για την ψυχική υγεία στο Βίλνιους 10 και 11 Οκτωβρίου του 2013. Τα σημαντικά θέματα των, ε, που αφορούν την ψυχική υγεία και κοινωνικά θέματα επίσης συζητήθηκαν και αναζητήθηκαν λύσεις το Φόρουμ Υγεία, βιώσιμα συστήματα υγεία για βιώσιμη ανάπτυξη θα γίνει στο Βίλνιους 19-20 ε, Νοεμβρίου όπου θα υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε για τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγεία. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σα ευχαριστώ για την ευγενική σα προσοχή. Ε, χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία να σα ενημερώσω για την πρόοδο τη Λιθουανική Προεδρία στον τομέα τη υγεία και να απαντήσω και στι ερωτήσει σα. Ε, έχουμε πολύ στενέ ε, σχέσει εργασία με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή ειδικότερα ε, και αυτό δημιούργησε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Προσβλέπω σε συνεργασία επικοδομητική για να προωθήσουμε το θεματολόγιο της υγείας και να ε, έχουμε μια πιο αποτελεσματική ε, πολιτική υγείας της Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes, of course we agree. And, uh, thank you very much for your presentation. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας γερμανικά επίσης σας ευχαριστώ πολύ, αλλά και για την καλή προετοιμασία. Και τώρα αρχίζουμε τον πρώτο γύρο, Γκροστέτ, Ροτ Μπέρεντ, Ρεμπέκα και Σοφία Κόνη. Η Φρανσουάζ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι συγγήτρια για το πρόγραμμα υγείας εδώ και ένα χρόνο προσπαθούμε να καταλήξουμε με τριμερή διάλογο, ο οποίος προβλέπεται για την Τετάρτη που μας έρχεται, με τους σκιώδεις εισηγητές βέβαια. Και συμφωνώ μαζί σας ότι το πρόγραμμα αυτό για την υγεία είναι θεμελιώδες. Άκουσα τι είπατε, είναι σημαντικό όντω να καταλήξει αυτή η υπόθεση, να ολοκληρωθεί. Τα κύρια σημεία σε κρεμότητα έχουν να κάνουν με το προπολογισμό, με το επίπεδο συγχρηματοδότηση των κοινών και με τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Ελπίζω να καταλήξουμε αυτή την Τετάρτη σε συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι ο προπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό υγεία διατηρείται. Για μα ήταν συνεκβάμων για να δεχτούμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το πρόγραμμα αυτό. Το συνολικό ποσό εξάλλου που προβλέπεται για το πρόγραμμα είναι 449 εκατομμύρια 394.000 ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Είναι μια αύξηση 394.000 σε σχέση με το αρχικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, στη σημερινή περίοδο είναι υπέροχο που καταφέραμε να πετύχουμε αυτή την μικρή έστω αύξηση. Αλλά για το επίπεδο συγχρηματοδότησης και της κατεξοδότηση πράξης, εδώ υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί εδώ μια λύση. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι η υγεία δεν πρέπει να είναι μια μεταβλητή ανάλογα με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό βασίζομαι στη Λιθουανική Προεδρία πραγματικά για να μας βοηθήσετε πραγματικά να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό την Τετάρτη και να βρούμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε για αυτά τα τεχνικά ζητήματα που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Η Ντάκμαρ Ροτμπέραντ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας και σας ευχαριστώ που τηρήσατε την υπόσχεσή σας να ξανάρθετε. Πραγματικά το εκτιμάω που προσπαθείτε να κάνετε τη διαφορά. Είναι πάντα δύσκολο να κάνει κανείς τη διαφορά. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Σας άκουσα προσεκτικά. Και όσον αφορά τους ιατρικούς εξοπλισμούς, Είπατε ότι θέλετε να πετύχετε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόοδο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό, γιατί το Κοινοβούλιο αποφάσισε στην γνωμοδότησή του για την πρώτη ανάγνωση πριν από δύο εβδομάδες και θεωρητικά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τους πρώτους τριμερείς διαλόγους. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε ακόμα μακριά από αυτό το στόχο. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι πρέπει να επιταχύνουμε αν θέλουμε αυτά τα δύο νομοθετήματα του κυρίου Λίζε και το δικό μου να προχωρήσουν. Συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη κάπως περισσότερο. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η ομάδα εργασίας ίσως αν δεν μπορεί να αποφασίσει πρέπει να παρακαθεί και να πάμε κατευθείαν στην Κορεπέρ και να γίνουν διαπραγματεύσεις πια σε πολιτικό επίπεδο. Σας άκουσα προσεκτικά και άκουσα τις φιλοδοξίες σας όσον αφορά τα τέλη που πρωτοσυζητάμε στην Επιτροπή μας. Και γιατί έχω αυτή την περίεργη αίσθηση στο στομάχι μου ότι για τον ιατρικό εξοπλισμό το βήμα θα μπορούσε να είναι πιο αργό, ενώ για τα τέλη τα κράτη-μέλη περιμένουν τα χρήματα να πηγαίνουν σε... στα ίδια. Δεν βλέπω εδώ να επιταχύνεται. Εντάξει, ξέρω ότι δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, αλλά ξέρω ότι ειλικρινά θέλετε να προχωρήσετε, αλλά βλέπετε είμαστε εσείς, εγώ και ο κύριος Λίζε. Δεν φτάνουμε. Μπορείτε να επηρεάσετε την ομάδα εργασίας και τους συναδέλφους σας στην ομάδα εργασίας. Μπορείτε να προσπαθήσετε παρακαλώ να πιέσετε και τους πρέσβεις στην Κορεπέρ. Αλλιώς θα χαθούν αυτές οι υποθέσεις. Ευχαριστώ Ρεμπέκα Τέιλορ και μετά η Σοφία Κονή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την κοινή θέση στην οποία καταλήξατε όσον αφορά τον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Έχω μερικές ερωτήσεις όμως σε σχέση με αυτό. Η πρώτη έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα. Γιατί η θέση του Συμβουλίου μιλάει για το, τις σε προδιαγραφές από αυτές που έχουν ε, νομές ΕΠΑ. και Αυστραλία. Αν χρειαζόταν ενημέρωση ήταν για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Οπότε ρωτάω την άποψή σας. Πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ελαστικότητα για να πλησιάσουμε περισσότερο στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ανάμεσα στο 64 και στο 99 υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όσον αφορά τώρα πάλι τις κλινικές δοκιμές, μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η πρόθεση του Συμβουλίου. Θα διατηρήσει τις δοκιμές αυτές χαμηλής επέμβασης, θα τις διατηρήσει. Και άλλη μια ερώτηση έχω για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Εδώ έχει γίνει πρόοδος. Μπορείτε όμως να μας πείτε περισσότερα σε σχέση με τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα, αυτά που περιέχουν νοικοτήνη, γιατί νομίζω ότι στο Συμβούλιο είναι διαφορετική η θέση τους. Ευχαριστούμε κυρία Τέιλορ, η Σοφή Οκονή και μετά η κυρία Γιανακουδάκη τελευταία. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη, πολύ γρήγορη. Τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Δεν έχω εμπλακεί άμεσα, αλλά έχω εμπλακεί πολύ ε, άμεσα αυτή την εβδομάδα συζητώντας με πάρα πολλούς ανθρώπους ε, σε σχέση με την οδηγία αυτή για το... και, και, και μου λένε ότι θα έπρεπε καταρχάς να εφαρμοστεί σωστά η ισχύουσα νομοθεσία για το κάπνισμα, πράγμα που δεν συμβαίνει σε κάποια κράτη-μέλη. Για τα τέλη που αναφέρατε, τώρα έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε για το σημείο αυτό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές θέσεις. Του Συμβουλίου, της Κομισιόν και φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο παίρνει ένα τρίτο δρόμο. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να το λύσουμε. Και το τρίτο σημείο, για μια ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα βλαστοκύτταρα, που συνέντεξα εγώ πριν από μερικούς μήνες και είπατε ότι θα δώσετε μια συνέχεια. Αναρωτιέμαι σε, ποια, σε ποιο σημείο των, ε, ε, των προτεραιοτήτων σας βρίσκεται αυτό. Συγγνώμη πριν που δεν είδα τη σωστή σειρά. Μέα κούλπα, η Σοφή Κονή τώρα. Σας συγχωρώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, για τα τσιγάρα και για την οδηγία για τον καπνό. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Κατά τις μετακινήσεις μου στα διάφορα μέρη, μπόρεσα να φωτογραφίσω ή e-cigarettes, ηλεκτρονικών τσιγάρων, που ε, λένε ότι τα τσιγάρα αυτά δεν ε, ε, βλάπτουν την δημόσια υγεία ούτε προκαλούν ρήπαση αλλά είναι κάτι που προωθεί την υγεία. Ε, πρέπει να ε, αντιδράσουμε στο μάρκετινγκ που σχετίζεται με τα τσιγάρα αυτά. Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με το σημείο αυτό, σε σχέση και με τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται ακόμη. Δεύτερο σημείο, που δεν είναι ε, κάτι το επίκαιρο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι επίκαιρο σε κάποια κράτη-μέλη σχετικά με τα ενεργειακά ποτά. Το Red Bull, παραδείγματο, για να φέρω μία μάρκα. Ποτά τα οποία καταναλώνουν σε μεγάλε ποσότητε οι νέοι μα σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ποτά που έχουν επίδραση πάνω στην υγεία, όπως ε, ο καπνός, το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθεσία για τα ενεργειακά αυτά ποτά. Στη Γαλλία φορολογούμε εδώ και λίγο καιρό τα ποτά αυτά για να τα κάνουμε πιο ακριβά ώστε να μην οθούνται να τα καταναλώνουν οι νέοι. Ε, Ποιος είναι ο προβληματισμός σας σε σχέση με τα προβλήματα αυτά που αύριο θα είναι πραγματικά προβλήματα δημόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προλάβουν ήδη από σήμερα και να αρχίσουν να συζητάνε αυτά τα προβλήματα. Φτάσαμε στο τέλος των παρεμβάσεων και ο Υπουργό έχει την τώρα τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις που έγιναν. Ορίστε. Αρχίζω με την πρώτη ερώτηση, το πρόγραμμα υγείας. Στις 6 Νοεμβρίου θα λύσουμε το θέμα οριστικά, εις ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό ε, και τα κοινά μέτρα και την, ε, τους συντελεστές συγχρηματοδότησης. Εγώ προσωπικά ε, νομίζω ότι αυτά τα 449 εκατομμύρια για την περίοδο 2014-2020 δεν φτάνουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όμως είναι προφανές ότι έπρεπε να συμφωνήσουμε. Διότι αυτά είναι αποτελέσματα συμβιβαστικών λύσεων που πρέπει να τα τηρήσουμε. Τώρα, οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα τεχνικά ζητήματα θα τα αντιμετωπίσουμε μέσα από εκτελεστικές πράξεις. Έτσι θα επιτελέσουμε την απαραίτητη πρόοδο. Εγώ είμαι εκπρόσωπος μιας χώρας φτωχότερης από τον ενωσιακό μέσον όρο, η οποία αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι και σε περιόδους οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπεται να γίνονται οικονομίες και να υπάρχει πολιτική λιτότητα σε βάρος του συστήματος υγείας. Και ευχαριστώ την ε, συνάδελφο Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ για την ερώτησή της. Τη συναντήσαμε, συζητήσαμε διμερώς ήδη για πολλά θέματα στον τομέα των ε, φαρμακευτικών προϊόντων δεν επιτύχαμε την ευκταία πρόοδο. Από την Ιρλανδική μέχρι τη δική μας Προεδρία, άμα δούμε τις εξελίξεις, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος στον τομέα των τελών. Όταν μιλάμε όμως για ασθενείς, ε, εκεί υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτά ε, σημαίνουν ότι ο κανονισμός ως νομοθετική πράξη ε, περιλαμβάνει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι δεσμευτικές λεπτομέρειες. Πρόκειται για αρμοδιότητες, για καθήκοντα που κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να ρίξουμε πολλές ιδέες, αλλά παράλληλα πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι λεπτομέρειες συχνά απαιτούν περισσότερο χρόνο. Εμείς όταν αναλάβαμε την Προεδρία στο, συζητήσαμε στο άτυπο συμβούλιο και ρώτησα τους συναδέλφους μου υπουργούς αν θέλουν να διαδηλώσουν την πολιτική τους βούληση ε, να επιτελέσουμε πιο, πολύ, πιο μεγάλη πρόοδο. Και πάντοτε συναντούσα τους συναδέλφους και στο ενδιάμεσο των συμβουλίων για να καταπιαστούμε με θέματα ε, ιατροφαρμακευτικών βοηθημάτων, τα διαγνωστικά in vitro. Αλλά καταλάβαμε ότι πρώτα έπρεπε να λύσουμε τα θεμελιώδη ζητήματα και μετά να πιάσουμε τις λεπτομέρειες. Προφανώς μου απαντούσαν πάντα ότι πρώτα θα πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητες. Α, υπήρχαν και άλλα κράτη-μέλη που έλεγαν ότι ε, θα εξέφραζαν επιφυλάξεις για διάφορους λόγους. Εμείς προσπαθούσαμε όμως να πιέζουμε αυτές τις χώρες ε, παίρναμε τηλέφωνο, ασκούσαμε πιέσεις, όλα αυτά πάντοτε για χάρη της πρόοδου. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξαναρχίσουν, ούτω ώστε να πάμε στην Κορεπέρ. Υπάρχουν θέματα που μπορεί να μην λύνονται στην ομάδα εργασίας. Εμείς πρέπει να δούμε πώς θα τα λύσουμε και πώς θα μπορέσουμε να ξαναδούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα όλο το κείμενο για να κινηθούμε και προς τα μπρος. Και στο Συμβούλιο καταγράφουμε τις θέσεις μας και βλέπουμε τι σχέση έχουν οι θέσει των κρατών μελών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί. Αυτή τη βδομάδα θα ξανακάνουμε συζήτηση και εγώ θα απευθύνω και επιστολή σε κάποια κράτη-μέλη και με τους 27 θα έρθω σε τηλεφωνική επικοινωνία. Μίλησα με τον Υπουργό, με τον Αρμόδιο Επίτροπο, με συγχωρείτε, σήμερα και ευχαρίστησα διότι μας επέτρεψαν να προσθέσουμε έναν αριθμό συνεδριάσεων. Δηλαδή θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να ε, υπάρξει πρόοδος το ταχύτερο δυνατόν. Και εις ό,τι με αφορά θέλω να είμαι ειλικρινής και δραστήριος, όσο γίνεται περισσότερο. Μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και επί Προεδρίας μας και μετά επί Ελληνικής Προεδρίας, αλλά οι επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Και εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε να καταφέρομαι αυτά που έχουμε θέσει ως στόχο. Τώρα, για τις ε, κλινικές δοκιμές. ε, απαντώ στη Ρεμπέκα Τέιλορ. Εκείνη, αν δεν κάνω λάθος, ρώτησε για τις κλινικές μελέτες και το χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό. Πρέπει να γίνουμε πιο ελκυστικοί σε σύγκριση με τους άλλους ανταγωνιστές μας, σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα πρέπει να γίνουμε πιο ελκυστικοί συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ε, σχεδιασμός των χρονοδιαγραμμάτων έχει να κάνει και με την προστασία των ασθενών, με την πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει, την τεχνογνωσία και με τα δικαιώματα των ασθενών. Γενικά τα δικαιώματα των ασθενών ε, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό και ε, ο σχεδιασμός των χρονοδιαγραμμάτων πρέπει να γίνει πολύ σωστά. Ε, αναφερθήκατε και στην οδηγία για τον καπνό και τη θέση του Συμβουλίου για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η κυρία Οκονή επίσης ρώτησε για αυτά. Στις ε, συζητήσεις με το Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Στη διαπραγματευτική διαδικασία αυτός ο κατάλογος είναι που έχουμε ε, καταρτήσει αποτελεί ένα θετικό βήμα παρόλο που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πολλές φορές και μεταξύ κρατών μελών. Εμείς πάμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Και εγώ ως γιατρός διαβεβαιώνω ότι έχω λάβει πάρα πολλές ε, επιστημονικές πληροφορίες που τεκμηριώνουν ότι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να είναι πλαβερό για την υγεία αυτά τα τσιγάρα μπορεί να τραβήξουν τους νέους που θα τα θεωρήσουν καλή εναλλακτική, αλλά η εξάρτηση από το ηλεκτρονικό τσιγάρο ε, είναι πολύ πιο κοντινή σε εκείνη από τα κανονικά τσιγάρα. Πάντως ε, διαφοροποιούνται λίγο εδώ τα κράτη-μέλη και πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση γιατί έχουμε το θετικό κατάλογο αφενός, αφετέρου έχουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και είναι σαφές ότι ο επόμενος τριμερής διάλογος θα είναι κρίσιμος. Πολύ σημαντικός. Και αυτό αυτές όλες τις ερωτήσεις πρέπει να τις απαντήσουμε κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Τώρα, δεν θυμάμαι ποιος έκανε την ερώτηση. Ε, πολλοί μπορεί να ισχυριστούν ότι δεν χρειαζόμαστε χωριστή οδηγία και ότι αρκούν τα συγκεκριμένα μέτρα. Αναφέρομαι εδώ στην οδηγία για τον καπνό αλλά εμείς ε, υπογράψαμε τη σύμβαση και δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, αυτά που αναλάβαμε να κάνουμε. Τώρα θα ασχοληθούμε με αυτά. Η οδηγία λοιπόν είναι ένα εργαλείο πολύ αποτελεσματικό. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν χρειαζόμαστε την οδηγία. Αυτοί που λένε ότι δεν χρειάζεται δεν καταλαβαίνουν τι αφορά. Από την άλλη, η καπνοβιομηχανία δεν θα είχε ασκήσει αυτή, αυτές τις τεράστιες πιέσεις αν δεν ήταν καθοριστική σημασία η οδηγία αυτή. Τώρα, για τα ενεργειακά ποτά. Και αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, το θέμα επίκαιρο στην ε, Λιθουανία αυτά τα ενεργειακά ποτά είναι πολύ διαδεδομένα μεταξύ παιδιών και εφήβων. Τα θέλουν, τα προτιμούν. Και υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ αυτών και της συνέχειας που είναι η κατανάλωση υνοπνευματοδών από τους νέους. Είναι λοιπόν αυτά ενεργειακά ε, ποτά τα οποία ε, μαστιγώνουν τον οργανισμό και μετά μπορεί κανείς να περάσει και στην κατανάλωση νοπνεύματος. Νομίζω ότι στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής σας υπάρχει και αυτό το θέμα που αφορά την ε, προστασία της υγείας. και έχει σχέση και με τις νόσους των νέων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικές οι συζητήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα και έχουν ε, λόγο ύπαρξης σε ορισμένες χώρες, κυρίως εκείνες όπου καταναλώνονται πολύ τα ενεργειακά ποτά. Τώρα, για τα βλαστοκύτταρα. Είναι κρίμα που κατά την Προεδρία μας δεν αφιερώσαμε χρόνο στη συζήτηση του θέματος αυτού. Στις ομάδες εργασίας ξέρουμε πολύ καλά τη σημασία του, του θέματος αυτού. Υπάρχουν πολύ προβληματικοί τομείς στην ιατρική ε, σε σχέση με το τα κύτταρα. Υπάρχουν δηλαδή πολλά θέματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Αλλά κατά την ε, Προεδρία μας ασχοληθήκαμε και με αυτό. Παρόλο που δεν ήταν στην ατζέντα της ε, Προεδρίας μας. Πάντως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων το συζήτησαν το θέμα των βλαστοκυτάρων. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι τα απάντησα όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γιατί ήταν διεξοδικότατες οι απαντήσεις σας και η ανακοίνωση ότι κάποια νομοθετήματα θα αντιμετωπιστούν θετικά από το Συμβούλιο είναι καλή. Γιατί πιέζει ο χρόνος, πλησιάζουμε στο τέλος της εντολής μας και ότι δεν προλάβουμε να το καταπιαστούμε θα σταματήσει, θα διακόπει. Αυτό είναι κρίμα. Κρίμα για την δουλειά που έγινε, κρίμα γιατί υπάρχουν πολλά θετικά που σημαίνουν προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό πασχίζουμε και συναντιόμαστε και ξανασυναντιόμαστε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε άλλη μια φορά και για να μας, να μας μιλήσετε ε, εδώ στην Επιτροπή. Σας εύχομαι και στο υπόλοιπο καλή επιτυχία. Λοιπόν, αύριο θα κάνουμε τις ε, ψηφοφορίες μας στις 10. Να φέρετε παρακαλώ όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες για την ψηφοφορία. Και καλωσορίζω και τον κύριο Κάστλερ προσωπικά που ήρθε σήμερα. Τον καλωσόρισα και στο Στρασβούργο και είναι τώρα το καινούριο πλήρες μέλος της Επιτροπής μας. Λύεται η συνεδρίαση, οι συντονιστές θα συνεχίσουν αύριο το πρωί στις 9 και όλοι οι άλλοι εξοπλισμένοι με τις ηλεκτρονικές κάρτες στις 10 η ώρα να έρθουν να ψηφίσουν. Καλό σας βράδυ.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

για